Uh, well, ladies and gentlemen, uh, we can get straight down to our business this afternoon. A very warm welcome. Να αρχίσουμε λοιπόν, λέει ο Πρόεδρος, απευθείας ε, τις εργασίες μας το απόγευμα. Χαίρομαι που βλέπω την αίθουσα τόσο γεμάτη τώρα που έχουμε μαζί μας ε, τον κύριο Επίτροπο, τον κύριο Μπαρνιέ. Όταν επιλέξαμε την ημερομηνία. Δεν γνωρίζαμε ότι θα είναι τόσο σημαντική ημέρα σήμερα και για την Κομισιόν και για την Επιτροπή μας, γιατί σήμερα, όπως ξέρετε, παρουσιάστηκε η οριστική ενιαία πράξη και λανσάρεται, δηλαδή παρουσιάζεται επισήμως και πιστεύω ότι θα έχει ορισμένες ερωτήσεις και μπορούμε οπωσδήποτε να υιοθετήσουμε το καινούριο σλόγγαν μαζί για τη νέα ανάπτυξη. Together for New Growth. Αυτή η φράση εκφράζει τις προσδοκίες μας και τις ε, προσλέψεις μας για ένα λαμπρότερο μέλλον πολύ ωραία και καλά. Χωρίς καθυστέρηση λοιπόν κύριε Επίτροπε θα ήθελα να σας δώσω το λόγο να μας μιλήσετε για την ε, κοινή αγορά αλλά και για τον ε, διαρθρωτικό για το δομημένο διάλογο και τα θέματα που εμπίπτουν σε αυτόν. Έχουμε ήδη εκμεταλλευτεί στο μέγιστο την παρουσία σας, έχουμε ε, συζητήσει πολλές φορές μαζί σας, αλλά τα θέματα είναι πολύ επίκαιρα και ενδιαφέροντα και θέλουμε να γνωρίζουμε τι φιλοδοξίες έχετε για το μέλλον, τι πιστεύετε ότι θα επιτύχει η ενιαία αγορά και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε στην περαιτέρω επιτυχία της. Όπως είπε και ο Λούις Γκρέχ, ε, η πρώτη, η πρώτη του έκθεση πριν από 11 μήνες επί του θέματος οδήγησε στη σημερινή κατάληξη και πιστεύω ότι οι διαμορφώνοντες την πολιτική στις Βρυξέλλες κινούνται με αργό ρυθμό. Όμως η ταχύτητα με την οποία εμείς μετακινηθήκαμε από ιδέες σε τελικές προτάσεις είναι ένα επίτευγμα σημαντικό. Πιστεύω ότι αυτό το αναγνωρίζετε και εμείς χαιρόμαστε ιδιαίτερα που, είμαστε, που έχουμε τη δική σας, το δικό σας, τα δικά σας φώτα σήμερα. Και σας δίνω το λόγο. Ε, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ Μάλκολ. Συγγνώμη για τη στενότητα χρόνου ε, διότι μετά από τη συνεδρίαση της ε, Κομισιόν σήμερα το πρωί, μετά από μήνες συζήτησης, εγκρίναμε την πρόταση για το Single Market Act, όπως επίσης και την ενισχυμένη συνεργασία για την Ευρωπαϊκή Ευρυσιτεχνία και την πρόταση του συναδέλφου μου του κυρίου Σεμέτα για την φορολόγηση της ενέργειας. Πρόκειται για μια πρόταση που αποτελεί έναν από τους μοχλούς του Single Market Act και σε λίγο πρέπει να πάρω και ένα αεροπλάνο για να πάω στη Στοκχόλμη που θα πρέπει να μιλήσω στο Σουηδικό Κοινοβούλιο για την τραπεζική κρίση. Πάντως ε, ευχαριστώ εξ αρχής ε, για την κατανόησή σας και κύριε, θέλω να ευχαριστήσω και τον πρόεδρο να πω κάτι προσωπικό για αυτόν. Ε, τον συνάντησα στο Στρασβούργο την ε, προηγούμενη εβδομάδα. Οι εκθέσεις Μπουσοτή, Κάμπος ε, και Κορέια συναντηθήκαμε με τον Μάλκομ είναι 11 επιτροπές οι οποίες εργάστηκαν με τη δική σας οστική δύναμη ε, ευχαριστώ τον Μάλκον ε, για την έκθεση ΕΓΕΣ ε, που έδωσε επίσης μια πνοή στην ενιαία αγορά. Δεν έχουμε βέβαια το, δεν παίζουμε τον ίδιο ρόλο. Και το έγγραφο που δημοσίευσε η Κομισιόν σήμερα το πρωί μπορεί να τύχει κριτικής, μπορεί μερικοί να μην είστε ικανοποιημένοι, άλλοι να μην βρουν αυτό που ήθελαν. Ε, όλα αυτά είναι λογικά. Πρόκειται για έναν δυναμικό συμβιβασμό μεταξύ των 27 επιτρόπων και εγώ ήμουνα πλάι στον πρόεδρο Μπαρόσο για να παρουσιάσουμε στον τύπο την ε, ε, ενιαία πράξη για την εσωτερική αγορά. Και πρέπει να πω ότι αν δεν ήσασταν εσείς παρόντες μέσα από τη διαφορετικότητα των πολιτικών ομάδων που αντιπροσωπεύετε, προτείνοντας, συζητώντας, ίσως να μην είχαμε καταλήξει εκεί που καταλήξαμε σήμερα. Σας ευχαριστώ ειλικρινά για την συνεργασία σας και τώρα πρέπει να δράσουμε. Πρόκειται για ένα framework, πρόκειται για έναν σιδηρόδρομο ε, θα σας ε, το εξηγήσω εντελώς τηλεγραφικά και θα σας εκφράσω και μερικές από τις πεπιθήσεις μου ως Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς. Πρώτον, τι θέλουμε εμείς για την Ευρώπη, θέλουμε να είμαστε θεατές ή πρωταγωνιστές στη διαμόρφωση του μέλλοντός μας. Όλοι το έχετε εδώ, ε, στο τραπέζι φαντάζομαι, εγώ ήμουνα στο Λονδίνο, μου δώσανε αυτό το τόσο καλογραμμένο έγγραφο και συγκινήθηκα γιατί κάπου αναφέρουν ε, και ένα δικό μου απόφθεγμα. Ε, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτός ο πίνακας, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και νομίζω ότι αποτελεί μια μείζωνα πολιτική έκκληση ε, δείχνει ότι άμα δεν προσέξουμε, άμα δεν πάρουμε τις σωστές αποφάσεις, όλα τα χρόνια, με τα χρόνια που θα περνάνε, εμείς ε, θα βγαίνουμε από την οθόνη του ραντάρ. Και για το 2050 από τις 10 πιο σημαντικές χώρες της Ευρώπης μόνο δύο θα είναι ευρωπαϊκές. Και θα συνεχιστεί το πράγμα έτσι. Θέλουμε να είμαστε λοιπόν πρωταγωνιστές ή θεατές. Εμείς θέλουμε να είμαστε πρωταγωνιστές. Και για να είμαστε πρωταγωνιστές η πρώτη βάση είναι η ενιαία αγορά. Δείτε τι γίνεται με τις Ηνωμένε Πολιτείες και την Κίνα. Η δεύτερη μου πεποίθηση είναι όπως εξάλλου συχνά το είπαμε αυτή η ενιαία αγορά δεν είναι όλη η Ευρώπη, δεν είναι όλες οι ευρωπαϊκές πολιτικές, είναι η βάση, είναι η πλατφόρμα. Αν αυτή η πλατφόρμα δουλεύει καλά, ό,τι και να βάλετε από πάνω, ιδιωτικές επιχειρήσεις, κυβερνήσεις, Ευρώπη, όλοι έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν καλύτερα. Και θέλουμε να λειτουργήσει σωστά. Τρίτη πεποίθηση Η Ευρώπη δεν πρέπει να είναι μόνο ε, μία γη κατανάλωσης. Δεν θα πρέπει να καταναλώνει μόνο τα προϊόντα που άλλοι παράγουν. Πρέπει να είναι μία, ένας χώρος παραγωγής ε, όπου θα παράγει τα δικά της αγαθά. Βρισκόμαστε σε μία φάση κρίσης οικολογικής, οικονομικής, οικολογικής, πολιτικής δεν θα βγούμε από την κρίση έτσι όπως είχαμε βγει πριν από 5-6 χρόνια. Η ανάπτυξη που θα ξαναφτιάξουμε πρέπει να είναι μια νέα ανάπτυξη. Αυτό το έλεγε ο πρόεδρός σας και αυτό είναι ένα σλόγγαν και πιο πολύ από όλους σλόγγαν. Όλοι μαζί για νέα ανάπτυξη, μαζί με τα κράτη-μέλη. Οι επαγγελματικές οργανώσεις, τα συνδικάτα, οι επιχειρήσεις, όλοι πρέπει να συνεργαστούμε για να δημιουργήσουμε μια νέα βάση και πιο ποιοτική βάση, πιο δίκαιη, πιο ανοιχτή. Εμείς εργαστήκαμε βασισμένοι στις 50 προτάσεις του Single Market Act για να βρούμε και όλες μας τις προτεραιότητες και οι προτάσεις που κάναμε είχαν ως στόχο να διαπιστώσουμε 12 τρόπους για να μπορέσουμε να βρούμε τους απαραίτητους ε, μοχλούς. Και για τον καθέναν από αυτούς ορίσαμε και μία δράση κλειδί, μία ουσιαστική δράση. Διότι είναι νέες, αποτελεσματικές για να λειτουργήσει πιο καλά η εσωτερική αγορά και σε δύο χρόνια αν υπάρχει πολιτική βούληση είναι λειτουργικές. Φτάνει να περάσουν από το Κοινοβούλιο και από το Συμβούλιο. Βέβαια δεν είναι αποκλειστικές αυτές οι 12 δράσεις κλειδί. Στο έγγραφο που θα διαβάσετε και σε έναν πίνακα που κάπου εδώ τον έχω, προσπαθώ να τον βρω τον πίνακα για τις 12 δράσεις κλειδί, οι στόχοι και μετά όλα τα συμπληρωματικά μέτρα που θα πρέπει να εφαρμοστούν παράλληλα οι συμπληρωματικές δράσεις με τη δράση κλειδί και συμβάλλουν αυτές οι συμπληρωματικές δράσεις στην επιτυχία της βασικής δράσης. Να σας αναφέρω τώρα αυτές που σας ενδιαφέρουν εσάς ως Επιτροπή ΙΜΚΟ. Λοιπόν, με τη σειρά. Χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσα από ένα ευρωπαϊκό διαβατήριο για, το, για τα κεφάλαια κινδύνου. Ένα ξαλάφρωμα των διοικητικών και λογιστικών ε, ε, βαρών των ΜΜΕ χορήγηση μιας επαγγελματικής ε, χάρτας και αναγνώριση των επαγγελματικών ειδικοτήτων, το, το, τα, τα δικαιώματα α, τα, ε, πνευματικής ιδιοκτησίας. Θα σας παρουσιαστεί το Μάιο μια γενική στρατηγική. Έχουμε μια συμβολική δράση. Ε, είναι το, η ευρυσιτεχνία και σήμερα προσέφερα εγώ στον κύριο Βαρόσο ένα έγγραφο το οποίο μου το στείλανε προχθές πρόκειται για μια από τις πρώτες εμπρισιτεχνίες στην Ευρώπη που είχε χορηγήσει το Ινστιτούτο Παστέρ για την κατασκευή της μπύρας. Το 1871 είναι αυτή η εμπρισιτεχνία. Και ο νέος τίτλος του Ευρω... της Ευρωπαϊκής Εμπρισιτεχνίας είναι 35 χρονών και εμείς σήμερα εγκρίναμε την δράση κλειδί για την εφαρμογή του μοχλού για την εύρηση τεχνία. Ελπίζουμε να κλείσουμε πριν από τα τέλη της χρονιάς με ενισχυμένη συνεργασία. Η Ισπανία και η Ιταλία οι οποίες είναι έξω από το χορό ελπίζω ότι και αυτές θα συμμετέχουν στην πρόταση. Έχουμε και άλλες τώρα συμπληρωματικές προτάσεις που θα σας παρουσιάσουμε σε επόμενες εβδομάδες. Συλλογική διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων, των ορφανών δικαιωμάτων, ε, εξυγχρονισμός της πολιτικής ε, της ε, πατέντας, ε, η καταπολέμηση της πειρατείας ε, και της απομίμησης. Η τέταρτη δράση είναι οι καταναλωτές και ο εναλλακτικό τρόπος επίλυσης των διαφορών και άλλες προτάσεις που αφορούν στους καταναλωτές, για παράδειγμα τα στεγαστικά δάνεια. Μετά έχουμε τις υπηρεσίες. Μιλάμε για εμπορικές υπηρεσίες. Η δράση κλειδί έχει να κάνει με την επέκταση της ε, ευρωπαϊκής εξομάλυσης της υπηρεσίας. Αυτό το ετοιμάζει ο κύριος Ταγιάννη για να αποφύγουμε τον κατακαιρματισμό των διατάξεων σχετικά με τις υπηρεσίες. Έχουμε δηλαδή διαφορετικές ε, διατάξεις πούμε, από τη μία χώρα στην άλλη για τις επιχειρήσεις καθαρισμού που τις εμποδίζει να πάνε να δουλέψουν από τη μία χώρα στην άλλη διότι υπάρχουν προβλήματα, για παράδειγμα πληροφορικού χαρακτήρα. Όταν εμείς μιλάμε για ευρωπαϊκή οικονομία υπηρεσιών, στις συμπληρωματικές δράσεις υπάρχουν θέματα ουσιαστικότατα. Πρέπει εμείς να εφαρμόσουμε τον μοχλό της οδηγίας για τις υπηρεσίες και αυτό το τονίζω κάθε φορά όταν πηγαίνω στις διάφορες πρωτεύουσες και συναντώ τους υπαλλήλου που έχουν αναλάβει να εφαρμόσουν αυτές τις οδηγίες. Και εγώ θέλω να αποδώσω όλη της, ε, την αποτελεσματικότητα σε αυτήν την ε, οδηγία. Μετά έχουμε τα B2B, έχουμε την ε, καταπολέμηση των αθεμήτων πρακτικών, ε, όλα αυτά δηλαδή που έχουν να κάνουν με τις ε, οικονομικές υπηρεσίες. Μετά έχουμε την ψηφιακή ενιαία αγορά. Εμείς θεωρήσαμε ότι θα πρέπει να διατηρήσουμε, να, να, να, να διασφαλίσουμε την ηλεκτρονική υπογραφή θέλουμε να έχουμε μία ομάδα για τα Trust Marks, δεσμευθήκαμε για αυτό το σχέδιο με εσάς. Έχουμε το θέμα της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο και τα δικαιώματα των καταναλωτών. Είναι ένα θέμα που έχει απασχολήσει ιδιαίτερα τον κύριο Ζουάπ. Για το θέμα της ε, κοινωνικής συνοχής εμείς ως ε, δράση κλειδί έχουμε ένα νέο μέσο που θα προτείνω σε μερικές ε, ε, εβδομάδες σχετικά με τα ταμεία αλληλεγγύης που θα διευκολύνουν τις επενδύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο και άλλα συμπληρωματικά μέτρα όπως το ευρωπαϊκό καθεστώς των Ιδρυμάτων ή το λάμπελ ε, περιηθικής ή οικονομίας αλληλεγγύης. Ο δέκατος ε, μοχλός είπαμε είναι ε, η συνοχή. Πρόκειται για την διευκρίνηση του τι καθολικές υπηρεσίες. Αυτό σας το είχαμε υποσχεθεί στο παρελθόν, όπως επίσης και η εφαρμογή του πακέτου ε, που, θα σας, που σας παρουσίασε ο συνάδελφος Αλμούνια. Δεν υπάρχει καμία αντίφαση μεταξύ εσωτερικής αγοράς και καθολικών ε, υπηρεσιών ε, υψηλής ποιότητας. Μετά έχουμε τις δημόσιες αγορές που θέλουμε να τις εξυγχρονίσουμε Έχουμε και το θέμα των παραχωρήσεων για την παροχή υπηρεσιών, ένα νέο πλαίσιο το οποίο σήμερα δεν υπάρχει. Μετά έχουμε το πώς θα διευκολύνουμε τη ζωή των μικρών επιχειρήσεων, κυρίως για σε λογιστικό επίπεδο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στην τελευταία στήλη του πίνακα, που δυστυχώς εμείς δεν έχουμε στην καμπίνα, εγώ δεν είμαι ο μόνος, όπως βλέπετε στον πίνακα, που έχει αναλάβει να προωθήσει αυτό το σχέδιο. Πρόκειται για ένα συλλογικό σχέδιο. Ο κύριος Μπαρόζο το υποστήριξε μέχρι τέλους. Ε, συνεχίστηκε η δουλειά του Μάριο Μόντι. Πάντως για αυτές τις 12 δράσεις κλειδί είμαστε τουλάχιστον 8 επίτροποι που δεσμευόμαστε από κοινού. 18 λοιπόν επίτροποι που θα ασχοληθούν μετά με τις συμπληρωματικές δράσεις. Σε αυτά δεσμευτήκαμε κύριε Πρόεδρε σήμερα το πρωί. Αυτό είναι το πλαίσιο δέσμευσης και τα σημεία κλειδί γύρω από το οποίο εμείς θα πρέπει να αποφασίσουμε. Να το ολοκληρώνω με κάτι το ουσιαστικό για αυτές τις 12 λειτουργικές δράσεις. Τις ανέφερα. Ευχαριστώ τη Σάντρα Καμίετε ε, για, το, για το θέμα της διακυβέρνησης εγώ δεν, δεν ανέφερα όλους τους, ε, τους μοχλούς πρόθεσης, ο κύριος Σεμέτα ασχολείται με αυτά. Πάντως ε, για την διακυβέρνηση, για να ολοκληρώνω, θέλουμε να εμπλέξουμε τους ε, πολίτες, είναι το Top 20 και το Φόρουμ της Ενιαίας Αγοράς, που θα γίνει στην Κρακοβία αυτό το πρώτο φόρουμ. αλλά θα ήθελα τα stakeholders, οι υπάλληλοι, τα συνδικάτα, οι επαγγελματικές οργανώσεις κλπ. να συναντιούνται τακτικά στην κάθε πρωτεύουσα, στην κάθε χώρα, να μπορούν να μαζεύονται, να έχουν ένα φόρουμ και να κάνουν τον απολογισμό. Εγώ προς στιγμή έχω κάνει ένα workshop ε, ε, σε 21 χώρες. Έχουμε μία δύναμη κρούσης, μία task force 600 υπαλλήλων σε όλες τις χώρες που ασχολούνται δηλαδή με τις ε, δημόσιες ε, με, τα, με τις ε, συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων κλπ. Και ξεκινάμε με αυτό τον πυρήνα των εθνικών υπαλλήλων και γύρω από αυτού θέλουμε να συσπυρώσουμε όλους τους οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους που ενδιαφέρονται για την εσωτερική αγορά, να αποκεντρώσουμε το τα φόρουμ αυτά σε κάθε χώρα. Εμείς θέλουμε να προσέξουμε πώς θα λειτουργήσουν αυτά τα αποκεντρωμένα ε, μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Έχουμε το iMile, ε, όπου θέλω του χρόνου να φτάσουμε σε 10 χιλιάδες του χρόνου. Το Σόλβικ αρχίζει και λειτουργεί καλά στην κάθε χώρα. Η Ευρώπη είναι δική σας, είναι κοντά σας. Θέλω όλα αυτά τα αποκεντρωμένα εργαλεία να λειτουργήσουν σωστά για να βοηθήσουν την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. εγώ είμαι έτοιμος με τους συναδέλφους μου να συνεργαστούμε με τους ε, μελλοντικούς εισηγητές. Ε, ε, με τρεις προεδρίες θα πρέπει να συνεργαστούμε. Πολωνική, Βανική και Κυπριακή μέχρι το τέλος του 2012 για να εργαστούμε εκ παραλίλου χωρίς βιασύνη. Θέλουμε να εργαστούμε κάπως πρωτότυπα για αυτές τις δράσεις κλειδί, όπως επίσης ε, και τα άλλα μέσα τα οποία σας ενδιαφέρουν, αλλά είναι, αποτελούν τμήμα των ε, συμπληρωματικών δράσεων. Αυτά για να σας πω έτσι στα γρήγορα το τι αποφασίσαμε σήμερα το πρωί. Uh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. μπορεί να μιλήσατε σύντομα, αλλά η έκθεση είναι πάρα πολύ πυκνή και γνωρίζουμε το περιεχόμενο. Βεβαίω, τονίσατε τα κεντρικά ζητήματα. Πολλοί συνάδελφοι θέλουν να μιλήσουν. Τεσσερισήμιση ώρα πρέπει να φύγετε, διότι πηγαίνετε στη Σουηδία, όπω είπατε. Έχω 16 στον κατάλογο, 17 τώρα. Και ο κ. Κόζιτσνεκ. Θα ήθελα λοιπόν να είσαστε πολύ σύντομοι και επί της ουσίας στις ερωτήσεις σας. Είμαστε τώρα 19 και αυξάνεται ο ρυθμός. Λοιπόν, καταρχάς, ε, ανά τρεις θα ακούσουμε τις ερωτήσεις για να απαντήσει ο Επίτροπος και πιστεύω ότι είναι. Καλή ιδέα να καλέσουμε τους εισηγητές της ε, πράξης της ενιαίας αγοράς ο κύριος Μπουζόη δυστυχώς δεν είναι εδώ, οπότε λέω να κάνουμε το εξής. Την κυρία Κανιέτη, Κορέντε Κάμπος και Γκρέχ επίσης να μιλήσουν, διότι είναι στην πρώτη γραμμή της ομάδας μας επί του θέματος. Να δώσω καταρχάς το λόγο σε εκείνους. Περιοριστείτε παρακαλώ σε ένα λεπτό. Εν συνεχεία θα έχω ένα γύρο ερωτήσεων από τους συντονιστές. Σβάμπ, Γκέπαρτ. Κρότσμαν, Μπίλε, Ρούλε και ο κύριος Τριανταφυλλίδης και μετά όλοι οι άλλοι. Θα προσπαθήσουμε να σας δώσουμε το λόγο ε, όσο πιο σύντομη τόσο καλύτερα. Είναι τώρα. Τέσσερις παρατέταρτο. Λοιπόν, είμαστε 22. Α, εξαρτάται τώρα με τη σειρά με τη σειρά όπως είπα. Πρώτα οι συντονιστέ και ε, όλοι οι άλλοι. Κυρία Κανιάτη, έχετε το, το λόγο. Έχετε ρολόι, ωραία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα κύριε Επίτροπε καταρχήν να σας συγχαρώ για την προσωπική σας δέσμευση υπέρ της εσωτερικής αγοράς. Τώρα όταν εγώ έριξα εδώ μια ματιά στις προτάσεις της Κομισιόν αυτοί και σε αυτούς τους 12 μοχλούς ήθελα πέρα από τους μοχλούς να μιλήσετε και για δέσμευση. Of the poetical leadership. Το μόνο που είδα είναι στην παράγραφο 5. η Κομισιόν θα παρουσιάσει προτάσεις στον νωρίτερο δυνατών για το καθένα από αυτά τα 12 σημεία ε, κλειδί. Χωρίς leadership, χωρίς ηγεσία δεν θα καταφέρουμε να, να δώσουμε μια πνοή, ένα ξεκίνημα στην εσωτερική αγορά. Αλλά και πάλι συγχαρητήρια παρόλα αυτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Πίτρο. Εγώ νομίζω ότι όλη αυτή η διεργασία ξεπέρασε τις προσδοκίες διότι έχουμε αυτόν τον κατάλογο των 12 που είναι πιο μικρό μικρός, πιο περιορισμένος κατάλογος από αυτό που είχαμε στην αρχή. Ο κατάλογος είναι πολύ καλύτερα οργανωμένος, αν μπορούμε βεβαίως να εκφραστούμε έτσι. Πέτυχε λοιπόν όλη αυτή η υπόθεση και χαίρομαι, εκφράζω την ικανοποίησή μου. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι. Η εισηγητές μας, όπως επίσης και οι σκιώδεις εισηγητές, αναγνωρίσαμε εδώ πέντε από τις βασικές μας ιδέες. Πέντε ιδέες μας βρίσκονται μεταξύ των 12 κατευθυντηρίων γραμμών που δίνεται των 12 μοχλών. Και το θέμα της απόσπασης των εργαζομένων το είχαμε χάσει κάπου και τώρα εδώ εμφανίζεται. Τώρα, για την αναγνώριση του ΣΥΓ του ΣΥ και του ΣΥΑΚ βλέπουμε απλώς να γίνεται μία αναγνώριση και χωρίς να γίνεται εγγύηση. Τώρα τι γίνεται όμως με την έρευνα. Γιατί η Κομισιόν δεν θα χρησιμοποιήσει τα Ροστάρις και τα ΡΕΚ που είναι πολύ σημαντικά ως εμπειρία. Και το χρήμα θα πρέπει να ακολουθεί την καινοτομία. Αυτά κύριε Επίτροπε. Είμαι πολύ επικής με τους εισηγητές, αλλά δεν θα είμαι τόσο επικής με τους άλλους. Ο Συμφωνώ, Πρόεδρε. Ο, στην εισήγησή του Επίτροπος κύριος Μπανιέ είπε ακριβώς τα εξής. Ότι χρειάζεται ηγεσία όλο αυτό το πλέγμα εργασιών για την ενιαία αγορά. Ηγεσία λοιπόν. Πολλές φορές έχω δηλώσει ότι δεν είμαστε βέβαιοι για το από πού προέρχεται η ηγεσία. Ένα τμήμα από το Συμβούλιο, ένα τμήμα από την Κομισιόν. Αλλά το περιεχόμενο των προσπαθειών είναι πάρα πολύ καλό. Χρειαζόμαστε όμως πολιτική ισχύ, πολιτική ηγεσία του Συμβουλίου. Του Συμβουλίου. Πιστεύετε ότι αυτή, αυτό το, το νέο ξεκίνημα θα είναι επιτυχές? Πριν απαντήσει ο κύριος Μπαρνιέ, θα ήθελα να χαιρετήσω την κυρία Πούσκας εκ μέρους της Ουγγρικής Προεδρίας και τον κύριο Σεφίλβαες ε, από την πλευρά της Επιτροπής. Ο ναι. κύριος Επίτροπος έχει το λόγο. Και εγώ θέλω να χαιρετήσω την αντιπροσωπεία της Ουγγρικής Προεδρίας, η οποία είναι ιδιαίτερα συνεργάσιμη και αλληλέγγυα σε όλη αυτή την υπόθεση. Να απαντήσω στον Λουιγκρέσο. το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπό την Προεδρία του κυρίου Ρομπόη αλλά και το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας υπό Ουγγρικής Προεδρίας και υπό Βελγικής προηγουμένως ε, συμμετείχαν σε όλη αυτή την υπόθεση. Εγώ έχω διαπιστώσει ότι για να ξεκινήσει μια πρωτοβουλία πρώτα πρέπει να ξεκινήσει από ψηλά, να αρχίσει να κατεβαίνει, να διαχέεται και μετά να ξανανεβαίνει. στην ιστοσελίδα μας είχαμε 840 ε, συμμετοχές, 840 παρατηρήσεις από πολίτες, ε, οργανώσεις, συνδικάτα ε, και είχαμε πάρα πολλές συζητήσεις με τους υπουργούς στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας αλλά και στο ΕΚΟΦΗΝ και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το Μάρτιο, μάρτυρα η Ουγγρική Προεδρία δώσανε μία όθηση στο Single Market Act. Ελπίζω δηλαδή ότι από το Ιούνιο και μετά μπορεί να έχουμε μια συλλογική δέσμευση στο πιο ψηλό επίπεδο. Πρόεδρος του Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της Ουγγρικής Προεδρίας, του Πρόεδρου της Κομισιόν για να μπορέσουμε πια να αποφασίζουμε. Και να απαντήσω στον κύριο Γκρέσ ο πρόεδρος, ο, ο κύριος από την αρχή υποστήριξε τις προσπάθειές μου. Εγώ θα ήμουν άδικος να, αν δεν έλεγα ότι χωρίς τον κύριο Γκρέσ θα είχα φτάσει εκεί που έφτασα. Να καταλήξουμε δηλαδή σε μια ομόφωνη ε, συμφωνία μετά από συμμετοχή όλου του σώματος ε, των επιτρόπων. Περάσαμε βέβαια μήνες για να αποφασίσουμε. Και το λέω στη Σάντρα Κανιέτε για τη leadership, για την αρχηγία. Βεβαίως ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του, αλλά ο καθένας μαζί με τους άλλους. Εμείς ε, πρέπει να αποφασίσουμε, άρα δεσμεύεται το σώμα. Και για τις 12 δράσεις κλειδί, εγώ είμαι αρμόδιος για τις 6. Και πολλοί από τους συναδέλφους μου για τις υπόλοιπες. Και μετά έχουμε ένα σωρό συμπληρωματικές δράσεις και θα δείτε ότι ορισμένε μπορεί να προχωράνε και πιο γρήγορα. Συμπληρωματικέ δράσεις δηλαδή θα προχωράνε πιο γρήγορα γιατί είναι πιο απλές, πιο όριμε από ότι οι δράσεις κλειδί. Δηλαδή το τελευταίο κομμάτι του Single Market Act που αφορά στην διακυβέρνηση, στη διαχείριση είναι κάτι το οποίο βασίζεται στις δικές σας προτάσεις. Και εκεί υπάρχει και η δέσμευση δηλαδή της Κομισιόν, το δικό της, ε, σε αυτό που της εμπίπτει δηλαδή τώρα και το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και αυτοί με τη σειρά τους πρέπει να δεσμευτούν και βέβαια ξέρετε ότι είναι υπέρ του γενικού συμφέροντος να δημιουργήσουμε σήμερα απασχόληση, να έχουμε καλύτερη διακυβέρνηση, να μειώσουμε τις δημόσιες δαπάνες, να έχουμε ρύθμιση, να έχουμε εποπτεία. Πρέπει να γίνουν όλα αυτά, όλες αυτές, όλοι αυτοί οι όροι είναι δύσκολοι όροι. Ε, και δεν μπορούμε να έχουμε ανάπτυξη και απασχόληση εύκολα χωρίς αυτούς. Τώρα για τον κύριο Κορέγια Ντεκάμπος, ε, για τις προτάσεις, είχαμε 50 προτάσεις ε, φυσικά και διαλέξαμε Αμερικές, μας είχε πει τότε το κοινοβούλιο ότι εδώ πρόκειται για ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο. Οπότε εμεί βγάλαμε αυτά τα 12, τους 12 μοχλούς που είναι λογική κινητικότητα, φορολόγηση, ε, ρυθμιστικό πλαίσιο, πνευματική διοκτησία. Τα βγάλαμε δηλαδή όλα αυτά, βρήκαμε τα πιο, ε, τα πιο ζούμερα για να διαπιστώσουμε, να δώσουμε τις προτάσεις. Ε, εσείς ε, για τις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος θεωρείτε ότι αυτή η πρόταση είναι ένα πρώτο βήμα. Μετά εσείς μπορείτε να εμπλουτίσετε τη συζήτηση, να τη συμπληρώσετε και για την πρώτη πρόταση κύριε Κορέια Ντεκάμπος για την έρευνα. βεβαίω συμφωνώ μαζί σας. Αυτό το οποίο προτείνουμε εδώ είναι το μέσο. δηλαδή το μέσο προς τα ποια κατεύθυνση πηγαίνει. Σίγουρα προτεραιότητα είναι η έρευνα και η καινοτομία για τις μικρές επιχειρήσεις. Αλλά εμείς τι θέλουμε. Θέλουμε ένα ευρωπαϊκό ε, μέσο για τα, για το κεφάλαιο κινδύνου και φυσικά μετά πρέπει να το προσανατολίσουμε προς την έρευνα, την καινοτομία. Ωραία, τώρα προχωρούμε στο γύρο των συντονιστών. Έχουμε μόνο το 35 λεπτά ακόμα και πάλι κάνω έκκληση να συντομεύετε. Ο κύριο Σφάμπ. Το πρωί μίλησα με την ταχύτητα του φωτό. Τώρα θα μιλήσω λοιπόν με μια πιο λογική ταχύτητα. Κύριε Επίτροπε, είπατε ότι η διαδικασία της εναέας αγοράς απέτησε ορισμένο χρόνο. Ναι, βεβαίως. Αλλά κατά τη διάρκεια αυτή πρέπει να προχωρήσουμε ε, συντονισμένα και θεσμικά και οριζόντια για να εξασφαλίσουμε την ε, ανάπτυξη. Ε, γι' αυτό ακριβώς πρέπει να προσέξουμε, να μην καθυστερούμε. Πολύ εμπλεκόμενοι είναι και ανυπόμονοι. Ο Μάριο Μόντι μας παρουσίασε ε, τα δεδομένα πέρσι και μας είπε πολύ σωστά ότι δεν χρειάζεται μόνο η οικονομική πτυχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και μία πτυχή και μία ε, αντιστοιχία με την εσωτερική αγορά. Πιστεύω λοιπόν ότι με την ενιαία αυτή η πράξη παρουσιάζεται μια μεγάλη ευκαιρία. Θα ήθελα να αναφερθώ σε τρία επιμέρους ε, σημεία. Καταρχάς θα πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στις ε, βασικές ε, δράσεις κλειδιά. Είναι όμως και άλλες συμπληρωματικές δράσεις που απαιτούν ταχεία εφαρμογή. Εκ μέρους του ΕΛΚ εμείς υποστηρίζουμε την προώθηση της δομοθεσίας με ε, δυναμικά, δηλαδή να προχωρήσουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα ε, το νομοθετικό πλαίσιο της ενέας αγοράς ε, μέσα στο 2000, μέχρι το 2012. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκέπχαρντ. Ευχαριστώ κύριε πίτροπε. Αναφερθήκατε στην ε, ανάλυση η οποία έγινε στο προηγούμενο βήμα, η οποία ανάλυση τόνισε ιδιαίτερα τις κοινωνικές ε, διαστάσεις ε, τα κοινωνικά ζητήματα που αποσχολούν τους πολίτες μας. Εγώ είμαι αρκετά απογοητευμένη διότι αυτή η θέση, αυτές οι ανησυχίες δεν αντανακλώνται στο έγγραφο αυτό το οποίο μας παρουσιάζεται σήμερα. Υπάρχει μεγάλο, μεγάλη ασάφεια και υπολείπεται κατά πολύ αυτών, αυτών των που αναμέναμε τουλάχιστον από πλευρά σοσιαλιστών δημοκρατών. Ωραία λέει μερικέ γενικότητε, εμβάθυνση στα κοινωνικά ζητήματα, αλλά δεν είναι ακριβώς αυτά που αναμέναμε ε, δεδομένου ότι οι πολίτες μας ανησυχούν ιδιαίτερα για το, το μέλλον, την ποιότητα ζωής. Αυτή η ανακοίνωση είπατε ότι θα παρουσιαστεί στο τέταρτο τρίμηνο, δηλαδή στο τέλος του χρόνου. Μα αυτό είναι πολύ αργά. Θα βοηθήσει αυτό στο να βρούμε λύση εντός του 2012. Πιστεύω ότι αντιτίθεται στην αρχική υπόσχεση που μας είχετε δώσει. Ο κύριος Κρότσμαν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πιστεύω ότι αυτά τα οποία έχετε επιτελέσει κύριε Πίτροπ είναι εξαιρετικά. Εξαιρετικά διότι ήταν πυκνά, συγκεντρωτικά και παρουσιάσετε ταυτόχρονα ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο μπορούμε να διευθετήσουμε φέτος. Θα, θα υπάρχει λοιπόν, ε, δίνει το χρονοδιάγραμμα ένα δυνατό έναυσμα, μια σπροξιά για να προχωρήσουμε με δυναμισμό. Αυτά τα 12 στοιχεία που παρουσιάσετε είναι κλειδιά, αλλά το πρώτο κλειδί είναι η διάθεση, η χορήγηση κεφαλαίου κινήσεως στις επιχειρήσεις και δι μικρομεσές. Οι μικρομεσές επιχειρήσεις είναι 12 εκατομμύρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν μπορεί κάθε μία να δημιουργήσει μία θέση εργασίας, τότε θα λύσουμε το πρόβλημα της ανεργίας. Το πιο δύσκολο πρόβλημα βεβαίω των επιχειρήσεων αυτών είναι η πρόσβαση στις, ε, στις αγορές ε, ε, παροχής κεφαλαίων κινήσεως έχουμε νομοθετικές προτάσεις και ε, παντού σε όλες τα 12 σημεία κλειδιά υπάρχουν ομοθετικές πτυχές. Θα σας παρακαλούσα κάνω μια έκκληση να προσέξετε ιδιαίτερα αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν για τους μικρομεσαίους και να προσέξετε ιδιαίτερα να μην τους επιβαρύνετε υπερβολικά με, κανονιστικό, με ένα κανονιστικό βαρύ πλαίσιο έτσι ώστε να μπορέσουν να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους στην εσωτερική αγορά. Ευχαριστώ πολύ ο Επίτροπος. Εμεί euh, eh. εμείς εδώ στην, στην αίθουσα με την ομάδα μου σημειώνουμε όλα όσα μας λέτε. Βέβαια υπάρχει, πρέπει να είμαι σύντομος ε, θα σας, μπορούμε να σας απαντήσουμε και γραπτός. Ο Ζουάμπ ανέφερε την οριζόντια και κάθε τη διαδικασία, τον ευχαριστώ. Εγώ νομίζω ότι η ποιότητα βέβαια θα πρέπει να πηγαίνει, να προηγείται της ταχύτητας. Γι' αυτό λοιπόν η επιλογή των ε, δράσεων κλειδί κράτησε χρόνο. Ε, θελήσαμε εμείς η Κομισιόν να παράγουμε ποιότητα, κυρίως νομική ποιότητα και διαλέξαμε αυτές τις δράσεις κλειδί ότι είναι απτές, είναι παραδόσιμες. Ας πούμε το Κοινοβούλιο είχε ζητήσει κάτι για την ψηφιακή αγορά σχετικά με το roaming. Ε, με την ε, κυρία Κρός εμείς ε, θελήσαμε να έχουμε την I-Authentification ε, ε, γιατί είναι κάτι το οποίο μπορεί να δοθεί πριν από το 2012. Το roaming ε, χρειάζεται κάποια συμπληρωματικές εργασίες με τις οποίες ασχολείται τώρα και κάναμε αυτή την, επιλογή. Εγώ συμφωνώ με όλο αυτό το διάβημα της διακυβέρνησης, της governance, της εσωτερικής αγοράς. Αν θέλουμε όμως το 2012 να έχουμε έτοιμο το σχέδιο θα πρέπει οι 8 άμεσα, πιο, πιο άμεσα ενδιαφερόμενοι επίτροποι να μπορέσουμε να συντονιστούμε με τους 14-15 συγητές από διάφορες επιτροπές, τους δικούς σας και άλλους. Και εδώ πρόκειται δηλαδή για συλλογική εργασία και οι τρεις προεδρίες θα πρέπει επίσης να δεσμευτούν σε αυτή τη διαδικασία διακυβέρνησης. Πρόκειται για μια τεράστια συζήτηση που έγινε ειλικρινά μέσα, στην, μέσα στο Σώμα των Επιτρόπων για την ανταγωνιστική κοινωνική αγορά. Ε, μην ανησυχείτε για το σε ποια θέση βρίσκεται η μία ή η άλλη πρόταση. Εκείνο που, είναι, που πρέπει να δείτε είναι το περιεχόμενο για, την κοινωνική, ε, ε, για το κοινωνικό σκέλος, ε, για την ε, για τους εργαζόμενους, τις αποσπάσεις των εργαζόμενων, για τις ε, δημόσιες υπηρεσίες, οι ανησυχίες που εκφράστηκαν από την ομάδα σας, ε, δεν έχει όμως μόνο η ομάδα σας την αποκλειστικότητα για την κοινωνική διάσταση. Εγώ και εγώ αισθάνομαι υπεύθυνο για όλες αυτές τις διαστάσεις. Όλα αυτά λοιπόν θα τα βρείτε και στην ανακοίνωση, κυρία Γεμπάχτα, ε, για την ε, ε, για, την, για το κοινωνικό κομμάτι υπάρχει η πρόταση Monty Cross που προθεί ο κύριος Σαλμούνια και τον υποστηρίζω εγώ όσον αφορά στις κρατικές ενισχύσεις, τις τοπικές υπηρεσίες και συνεργαζόμαστε για αυτήν την ανακοίνωση που θα πρέπει να ε, ξεκαθαρίσει τα πράγματα για τις καθολικές υπηρεσίες. Αν κάνουμε την ανακοίνωσή μας στα τέλη της χρονιάς μπορεί να γίνει λειτουργική πολύ, πολύ γρήγορα. Κύριε Κρότσμαν, ευχαριστώ πολύ για την ε, υποστήριξή σας. 20 εκατομμύρια μικρές επιχειρήσεις για την πρόσβαση χρηματοδότηση των ΜΜΕ, για τις ε, δημόσιες αγορές, για τις δημοπρασίες και όλα αυτά. Όλα δεν θέλουμε εμείς να μπερδέψουμε τα πράγματα και ίσως ε, τα μπερδέψαμε πολύ στο παρελθόν. Δηλαδή πολλές μικρές επιχειρήσεις έχουν την αίσθηση ότι αυτή η μεγάλη αγορά δεν είναι φτιαγμένη για, για, για αυτούς. Ε. Είναι περισσότερο μία αγορά δεσμεύσεων και υποχρεώσεων ε, θέλουμε να ξαλαφρώσουμε κατά συνέπεια τους λογιστικούς ε, κανόνες, ε, τους διοικητικούς κανόνες, ούτως ώστε οι μικρές επιχειρήσεις να διαμορφώσουν την, ε, την αίσθηση ότι τέλος πάντων η Ευρώπη γίνεται κάτι το απλούστερο και διευκολύνει τις ανταλλαγές και τις εξαγωγές. Λοιπόν, προχωρήσαμε στον κατάλογο των ομιλητών, να συνεχίσουμε. Θα κάνουμε τους υπόλοιπους συντονιστές σε ομάδες των τριών, κύριος Μπίλαν, Ρούλα και ο κύριος Τριανταφυλλίδης και κατόπιν θα περάσω στις ομάδες των τεσσάρων. Κύριος Ρόσφορτ, ε, κύριε Ρόσφορτ και λοιπά. Λοιπόν, ετοιμάστε τις ερωτήσεις σας εντός στην πορεία και θα ξεκινήσουμε από τον κύριο Μπίλαν. Λοιπόν, θέλω να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που βρήκε χρόνο ο Επίτροπος να έρθει στην Επιτροπή μας την ίδια μέρα που δημοσιεύτηκε το σημαντικό αυτό έγγραφο. Το πρώτο έγγραφο αφορά το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας. Το περιμέναμε επί χρόνια και είμαι πολύ ικανοποιημένο. Αρχικά είχα εντυπωσιαστεί από τη μείωση του διοικητικού κόστους από πάνω από 30.000 σε κάτω από 700 ευρώ που βεβαίως θα κάνει τα διπλώματα αυτά πολύ πιο ανταγωνιστικά σε σχέση με τα αντίστοιχα των ΗΠΑ. Ως εκπρόσωπος μιας χώρας η οποία δεν θα ε, βλέπει τη γλώσσα της να εντάσσεται στις επίσημες χώρες, ε, χαίρομαι που θα ε, καλύπτεται το κόστος μετάφρασης. Τώρα, έχω μία ερώτηση για το έγγραφο της ενιαίας αγοράς. Μπορείτε να μας πείτε κάτι με τους, τους δύο πρώτους μοχλούς. Πρώτον, η βελτίωση της προσβασιμότητας στις χρηματοπιστωτικές αγορές για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και δεύτερον, η αυξημένη ε, κινητικότητα των εργαζομένων. Μήπως μπορείτε να γίνετε πιο συγκεκριμένος για την αμοιβαία αναγνώριση της οδηγίας των ε, ε, επαγγελματικών προσόντων. Ευχαριστώ. Κύριε Ρίλε, σας ευχαριστώ που ήρθατε σήμερα, κύριε Επίτροπη κύριε Επίτροπε, διότι είναι πολύ σωστό να συμμετάσχουμε στην διαδικασία από τις πρώτες φάσεις, τα πρώτα βήματα. Υποστηρίζονται περισσότερα από αυτά που είπατε. Βεβαίως είπατε ότι η νομοθεσία ε, πρέπει να οδηγήσει σε βελτίωση της νομοθετικής ποιότητας θα πρέπει να βοηθήσει η νομοθεσία την νομική διαφάνεια, την νομική ασφάλεια και να μην δημιουργήσει νομικές ασάφειες, ιδίω για τις μικρομεσαίες. Ε, αυτό που σημείωσα για τις συμπληρωματικέ δράσεις είναι η αηφορία, ε, το περιβάλλον, ε, πράσινη οικονομία. Στην πατρίδα μου και στο κρατήδιό μου, στη Βάδη Βιρτεμβέργη, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι πολύ καινοτομικέ. Ε, ιδιαίτερα στην πράσινη πτυχή. Χρειάζονται όμως ενίσχυση ευρωπαϊκή. Και στο θέμα της ενέργειας, ε, της ε, μείωσης της εξοικονόμησης ενέργειας και άλλων πράσινων μέτρων έχουν πολύ καλά παραδείγματα. Ο κύριος Τριανταφυλλίδης. Θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί όπως σας είπα και στο Στρασβούργο κάνετε πάντοτε τις ομιλίες σας πάρα πολύ ενδιαφέρουσες και μας κρατάνε σε εγρήγορση. Ενδιαφέρουσες είναι και οι δράσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό το φυλάδιο παρόλο που δεν βλέπω τίποτα για τα τυχερά παιχνίδια παρότι ήταν μέσα στις προθέσεις της Επιτροπής να θίξει αυτό το θέμα. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω συγκεκριμένα προτίθεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει σε ρύθμιση της κοινοτική νομοθεσίας περί τυχερών παιχνιδιών ώστε να ρυθμίζεται πανευρωπαϊκά ο κλάδος και ποιες οι σκέψεις και οι επιθυμίες της Επιτροπής για ένα τέτοιο ευαίσθητο θέμα δεδομένου ότι μέχρι στιγμής υπάρχει ισχυρή προστασία για τις εθνικές διατάξεις κάτι άλλωστε που έχει συμπεριληφθεί σε σειρά αποφάσεων του ΔΕΚ για την δυνατότητα των κρατών μελών να διατηρούν περιοριστικές διατάξεις. Ευχαριστώ πολύ. Thank Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας για τις πολύ ε, συγκεκριμένες ερωτήσεις σας. Κύριε Βίλαντ, σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια για τις ευρυσιτεχνίες. Εγώ θα είμαι απόλυτα ικανοποιημένος και να είμαι ειλικρινής μόνο όταν η Ισπανία και η Ιταλία ενταχθούν στην πρόταση που θεωρώ ότι είναι οικονομικά ζωτική και απολύτως απαραίτητη για τις επιχειρήσεις, κυρίως τις μικρές και πολιτικώς αποδεκτή για όλες τις κυβερνήσεις πολιτικός αποδεκτή και οικονομικός απαραίτητη. Ελπίζω και μετά σας διαβεβαιώ ότι θα έχουμε, παρουσιάσουμε το Μάιο ένα νέο κείμενο για την νομοθετική δομή που θα χρειαστεί να, για να συνοδεύσουμε αυτόν τον ενιαίο τίτλο προστασίας. Και αυτό βάσει της πρόσφατης απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Τώρα δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες για το τι θα κάνουμε για να ευκολύνουμε τη χρηματοδότηση των ΜΜΕ. Υπάρχει αυτή η ιδέα να δούμε αν μπορέσουμε δηλαδή ορισμένες πιστώσεις ε, ε, στον τομέα των κεφαλαίων κινδύνου όπως επίσης ε, μου έχει περάσει από το νου μια πρόταση για ένα ευρωπαϊκό χρηματιστήριο για τις ΜΜΕ περιφερειακές, περιφερειακά ή εθνικά χρηματιστήρια. Ας πούμε, στη Γερμανία, για παράδειγμα, υπάρχουν μερικές ειδικέ διαδικασίες και μερικά ειδικά προϊόντα που επιτρέπουν ε, την πρόσβαση των μικρών επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση. Αλλά ε, και λόγω του ενδιαφέροντός σας, ε, κύριε Βίλαντ, για αυτό το θέμα θα σας πληροφορώ τακτικά σχετικά. Κυρία μου, χωρίς να είμαι πράσινος, εδώ και πάρα πολύ καιρό έχω δεσμευτεί για, στον τομέα αυτής της νέας ανάπτυξης. Γι' αυτό εγώ ήθελα να ε, όλοι μαζί για τη νέα ανάπτυξη, new growth. Εγώ επένδυσα σε αυτό το σλόγγαν διότι ήθελα ε, να, έχουμε και αυτή τη διάσταση μέσα στο growth, στο new growth. Εγώ υποστηρίζω τις ιδέες ε, που βοηθούν να διαμορφώνεται ένα αίσθημα ισότητας μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών που ακόμη δεν είναι τόσο στέρεο. Και εγώ ε, δρώ ούτως ώστε τα μπόνους που πληρώνουν οι τράπεζες να μην φτάνουν σε αυτά τα ανεξήγητα και αδικαιολόγητα ε, ύψη όταν 10% των Ευρωπαίων είναι άνεργοι και τόσες ε, χώρες απαιτούν πια τόσες προσπάθειες από τους πολίτες τους. Περισσότερη ισότητα λοιπόν δικαιοσύνη και ε, πράσινη αηφόρα ανάπτυξη. Δείτε ε, τις ε, προτάσεις κλειδί. Πολλές από αυτές τις προτάσεις αφορούν τα δικά σας ε, ενδιαφέροντα. Δείτε την πρόταση του κυρίου Σεμέτα για τη φορολόγηση της ενέργειας που στη χώρα σας συζητιέται πολύ. Αυτό έχει να κάνει όμως συνδέεται με την αποτελεσματικότητα του φορολογικού συστήματος για να πετύχουμε μια νέα ανάπτυξη. Οι δημόσιες υπηρεσίες, ο εξυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων υπηρεσιών, και ε, και μάλιστα πριν γίνω επίτροπος ε, για τις... Ε, α, συγγνώμη, για τις δημόσιες αγορές, ε, όχι, όχι τις, τις δημόσιες υπηρεσίες, έκανα λάθος, λέει ο επίτροπος, για τις... για τις κρατικές προμήθειες, για τις δημοπρασίες, τους εντολοδόχους κλπ. που θέλουν, θα, ενισχύουμε αυτούς οι οποίοι θέλουν να ενισχύουν την απασχόληση, ε, το, δεν, κάνουν αποκλεισμούς, ε, προωθούν την αηφορία. Ξέρουμε επίση ότι η απασχόληση κρύβεται και στις νέες τεχνολογίες, στο περιβάλλον. Ξέρουμε επίση ότι έχουμε τις εμπρισσοτεχνίε, την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησία και και και στο θέμα της ποιότητας της ανάπτυξης όλα αυτά παίζουν ένα ρόλο. Μεταξύ των γραμμάτων μπορείτε να δείτε διάφορα θέματα τα οποία ενηχεύουν και επηρεάζουν την ανάπτυξη με διαφορετικό τρόπο. εγώ εδώ και καιρό... Ε, εδώ και καιρό με απασχολεί το θέμα ότι το περιβάλλον δεν είναι κάτι το οποίο το έχουμε έτσι πρέπει να το αφήσουμε στις επόμενες γενιές. Κύριε Τρενταφυλλίδη, βεβαίως και πρέπει να δράσουμε επί του τζόγου. Διότι περνάνε πάρα πολλά χρήματα από εκεί μέσα. Εγώ ε, ε, ξεκίνησα ε, μια πράσινη βίβλο πριν από μερικές μέρες. Και είμαστε έτοιμοι να ανασύρουμε όλα τα διδάγματα από αυτήν την πράσινη βίβλο για να μπορέσουμε να διαφυλάξουμε και μερικά ουσιαστικά θέματα κοινωνικά, δηλαδή η προστασία ε, των ανηλίκων, ε, λεύκανση χρήματος, εθισμός, ε, και άλλα κοινωνικά φαινόμενα που προκύπτουν. Λοιπόν, κυρία Ρούλερ είναι η συγγήτρια για τις κρατικές προμήθειες, τις οποίες θα συζητήσουμε σύντομα. Έχουμε τρεις ομάδες των τεσσάρων. Πρώτη ομάδα, ο κύριος Ρόσφορτ, Κρόσπερ, Βάνιου και ο κύριος Μάντας. Και μετά το Μπούσετιλ, Βάιλαρ, Αριάς και Λεγκρίπ. Και σας παρακαλώ, μία ερώτηση ο καθένας για να τα καταφέρουμε. Ο κύριος Ρόσφορ, το ένα λεπτό σας. Μπράβο, μπράβο κύριε Επίτροπε, σας υποστηρίζουμε ιδιαίτερα δυναμικά. Τώρα αυτός ο Βρετανικός πίνακας που μας δείξατε προ λίγο, μα τη λύση την ξέρουμε πολύ καλά. Κάποια στιγμή πρέπει να έχουμε και ένα τετραγωνάκι που θα γράφει Ευρωπαϊκή Ένωση Εκεί όμως δεν έχουμε φτάσει ακόμα. Και όταν θα φτάσουμε όμως εκεί θα είμαστε μεταξύ των top 3. Σήμερα είμαστε μπροστά από την Κίνα, αλλά σε μερικά χρόνια δεν θα είμαστε. Και γιατί σας τα λέω αυτά. Διότι εγώ θεωρώ ότι αυτή η νέα ανάπτυξη που ανακαλύψαμε είναι ένα στη εσωτερικής ανάπτυξης στην εσωτερική αγορά αλλά και ανταγωνιστικότητας έναντι του, του υπολείπου κόσμου. Ξέρω ότι είναι πάντα εύκολο να κάνει κανείς κριτική, αλλά θεωρώ ότι 12, αυτά τα 12 μέσα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Δεν είναι όμως επαρκή για να έχουμε ε, μία εκτόξευση προς τον υπόλοιπο κόσμο. Ας πούμε, 21ος αιώνας επένδυση στα, στα καθαρά αυτοκίνητα που θα μπορούν να εξάγονται, ε, χίλια δυο πράγματα, τι κάνετε εσείς ε, για να προσανατολίσετε αυτή την ανάπτυξη, ούτως ώστε να μπορέσουμε να αναπτυχθούμε και προς τα έξω. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι πρόκειται για μια μεγάλη μέρα για την Ευρώπη. Χάρη νημών κύριε Επίτροπε. Έχουμε πλέον κάτι το συγκεκριμένο για να προχωρήσουμε και να ολοκληρώνουμε την εσωτερική αγορά. Κυρίως για να υποστηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το ηλεκτρονικό εμπόριο και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Υποστηρίζω όλες τις προτεραιότητες που υποδείξατε. Για το εμπόριο θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που λάβατε υπόψη σας ε, την δική μας άποψη για την ανάληψη πρωτοβουλειών για τις εμπορικές πρακτικές. Και ρωτώ, πώς αντιμετωπίζετε αυτό το γενικότερο πλαίσιο για την αναζωγόνηση του ευρωπαϊκού εμπορίου. Εγώ το έχω συμπεριλάβει βέβαια στην έκθεσή μου για το εμπόριο και έχει μία, ένα μακροπρόθεσμο όραμα για να μπουν στην ημερήσια διάταξη της Ευρώπης όλα τα ζητήματα που αφορούν στο εμπόριο. Τα goods package, η κίνηση, των διακίνηση αγαθών, ευρωπαϊκό σύστημα πληρωμών κλπ. Τι θα κάνετε και αυτά για να τα σμπρώξετε. Ένα λεπτό 22 δευτερόλεπτα κύριε Πρόεδρε πολύ καλά. Ε? Ναι, αλλά για τρεις ερωτήσεις, <laughs> κύριε Βενιούρ. Εγώ θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομη. Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ που το παρουσιάσατε το κείμενο, αλλά και για τη μέθοδο πρόκειται για κάτι το πρωτότυπο και σπάνιο, θέλω να το τονίσω αυτό. Μιλήσαμε εδώ για ηγεσία, ότι η, εσωτερική, ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά πρέπει να τραβήξει την παγκοσμιοποίηση προς τα πάνω, διότι είναι και η πρώτη αγορά παγκοσμίω και πρέπει να βρούμε από κοινού μία στρατηγική για τον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Εγκρίνω απόλυτα όλα όσα γράψατε και για την επαγγελματική εξειδικευσή, την πνευματική διοκτησία, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τις ε, δημοπρασίες, κρατικές προμήθειες, ε, και το είναι βρυσή τεχνία. Αλλά κάπου κάτι με, με, ενοχλεί. Γιατί για να μπορέσει κανείς να δώσει κίνητρο σε μια πραγματική ανάπτυξη πρέπει να δημιουργήσει και πραγματική απασχόληση. Βιομηχανική απασχόληση η οποία επιπλέον να σέβεται και το περιβάλλον δεν γίνεται χωρίς εργαζόμενους και στις ε, προτάσεις που κάνετε εσείς για την εγγυήση των κοινωνικών δικαιωμάτων των εργαζομένων, ας πούμε για τους αποσπασμένους εργαζόμενους, στο 10 για την ανακοίνωση, για τις κοινωνικές υπηρεσίες καθολικού συμφέροντος και ε, τις δημόσιες υπηρεσίες καθολικού συμφέροντος, σε πραγματικά κάτι μου λείπει. Μένω με την όρεξη. Βέβαια, κάνετε και ένα ενδιαφέρον σαρδάμο μιλώντας ε, και με το σαρδάμ που κάνατε κάπου εγώ κρατάω την ε, ε, ευελπιστώ. Θα έχω ένα πρόβλημα, ένα πρόβλημα. Γιατί εγώ στις 5.30 έχω ένα αεροπλάνο για τη Στοχόλμη Και να ξανάρθω άμα θέλετε, μια άλλη φορά δηλαδή, για να πω... Κύριε Ροσφόρ, κύριε Ροσφόρ. Και κυρία Βερνιούκ, σας ευχαριστώ. Το Single Market δεν είναι όλη η Ευρώπη και όλες οι ευρωπαϊκές πολιτικές. Για πλατφόρμα μιλάμε. Για βάση της οικονομίας. Πρέπει να λειτουργεί εύρυθμα. Από πάνω έχουμε ένα σώρο πολιτική που πρέπει να φτιάξουμε. Ιδιωτικέ και δημόσιες πρωτοβουλίες. Για να μπορέσουμε να προσανατολίσουμε την Ευρώπη προς μια οικονομική και κοινωνική κατεύθυνση. Για να λειτουργήσει καλά η εσωτερική αγορά. Και το πρώτο πράγμα για μένα είναι η ευρυσιτεχνία βρίσκεται στη βάση του Single Market Act. Αν δεν έχουμε ευρυσιτεχνία τότε εμεί επιβαρύνουμε όλες μας τις επιχειρήσεις έναντι των Αμερικάνων και των υπόλοιπων. Δεν τις βοηθάμε. Μπαίνουν ένα σωρό προϊόντα μαϊμούδες στην αγορά. Κακά προϊόντα για τη δημόσια υγεία που καταστρέφουν και 200.000 ε, θέσεις εργασίας το χρόνο. Επίσης, οι ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις για την έρευνα και την τεχνολογική και, την καινοτομία θα είναι πιο αποτελεσματικές. Βάση είναι το, το ΣΜΑ. Δεν είναι ε, πολιτική. Είναι βάση για πολιτικές. Κύριε Ροσφόρ για την ανάπτυξη εσωτερική, εξωτερική. Εμείς ε, σαφώς και έχουμε κατά νου την εξωτερική ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς και με τον συνάδελφο Ντεγκούχτ θα προτείνουμε εντό των ημερών ε, το θέμα της συμφωνίας GPU ε, ε, για τις χώρες εκείνες οι οποίες δεν κάνουν τίποτα ως προς την αρχή της αμοιβαιότητας, ενώ εμείς την κρατάμε δηλαδή την αμοιβαιότητα απέναντί τους, αυτοί μένουν απαθείς. Τώρα κύριε Σβάμπ, αυτό που είπατε είναι πολύ σημαντικό. Εγώ πριν από το τέλος του καλοκαιριού θα παρουσιάσω το σχέδιο δράσης ε, για το εμπόριο και θα συμπεριλαμβάνονται και πολλές από τις προσατάσεις σας για νομοθετικά μέτρα. Θα κρατήσουμε και το ευρωπαϊκό σύστημα πληρωμών, θα το προχωρήσουμε ε, και για την οδηγία του ηλεκτρονικού εμπορίου, του e-commerce. Με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα οι αθέμητες εμπορικές πρακτικές, ε, όπως επίσης και η σχέση μέσα στο δίκαιο εμπόριο, για ε, την στενή για, ε, επαφή αγοραστή-πολιτή. Κύριε Βερνιούκ, υπάρχουν πάρα πολλές προτάσεις οι οποίες ε, είτε είναι παρκής είτε όχι έχουμε την οδηγία για τους εργαζόμενους λοιπά. Σας ευχαριστώ που προσέξατε και στην πολιτική εισαγωγή του Single Market Art. Είπα στην κυρία Κανέιτε ότι πρέπει να είναι προσεκτική σε αυτά που είπαμε στην αρχή. Κοιτάστε, το σώμα των επιτρόπων τον έκρινε όλο αυτό. Υπάρχει δηλαδή μια συλλογική δέσμευση γύρω από αυτό. όπως έγινε και στο παρελθόν για την οδηγία υπηρεσιών. Κυρίε και κύριοι, έχει σχεδόν λήξει ο χρόνο. Κάνω μια προσφορά στου υπόλοιπου 8. Μπορείτε ο καθένα σε 30 δευτερόλεπτα να κάνετε μια γρήγορη ερώτηση. Πολύ ωραία, συμφωνήσαμε. Κύριε Μπούστομ, κύριε Βάλερ, κύριο Άρια, κύριε Λεγκρίπ, Κώση Νίκ. Κύριε Μάντε, κάτι χάσατε. Α, φταίει. Δεν είμαι συνηθισμένο. Ε, λοιπόν, μια ερώτηση προ τον Επίτροπο ένα πρόγραμμα δράσης, τα στηρίζω όλα, σας υποστηρίζω, αλλά πώς θα ε, γίνουν γνωστά όλα τα καλά πράγματα που κάνουμε στους ε, Ευρωπαίους πολίτες και να μην τους περνάνε ε, πάνω από το κεφάλι τους. Εγώ θέλω να μπουν μέσα στο μυαλό τους, όχι να φεύγουν. Έχετε σκοπό να προτείνετε ένα πρόγραμμα δράση από αυτού. Κύριος Μπρίζδερ. Euh, Κύριε Επίτροπε, η ερώτησή μου αφορά στη διεθνοποίηση των ΜΜΕ. Μόνο το 12% των ΜΜΕ δεσμεύονται σε διασυνοριακές δραστηριότητες. Και αν δεν ανοίξουμε την πόρτα ούτως ώστε οι ΜΜΕ να βγουν από τα εθνικά σύνορα, τότε πραγματικά δεν πετύχαμε τίποτα. Θα, παρα, ρωτούσα λοιπόν. Ποιο θα είναι το κερδίζον χαρτί στον τομέα της ε, διεθνοποίησης. Η κυρία Βάιλερ. Δύο πολύ σύντομα χάσα συγχαίρω για τη δέσμευση που δείξατε και το, το 10 κλειδί, η δράση την οποία περιμένω χρόνια και χρόνια. Τον Οκτώβριο ε, λάβαμε ορισμένες θαυμάσιες προτάσεις από εσά, 12 λάβαμε σήμερα. Σε δύο μήνες λίγη νομοθετική περίοδο της θητείας μας και δεν πιστεύω ότι η εσωτερική αγορά δεν θα προλάβει να αναζωογονηθεί μέσα σε αυτό το διάστημα. Κύριο Σαρίας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το Forest Research Center για το ηλεκτρονικό εμπόριο στη ΣΥΠΑ αναφέρει ότι το e-commerce είναι το αντιπροσωπεύει το 12,5% του συνολικού τζίρου του ηλεκτρονικού εμπορίου, του λιανικού συγγνώμη, εμπορίου στην ε, Αμερική. Και θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο για το 2015. Θέλω να ξέρω το σχέδιο δράσης το, για, το e-market ε, έτσι όπως παρουσιάζεται στο ΣΜΑ πώς ε, το έχετε κατά νου. Γιατί, εμείς έχουμε, γιατί έχουμε μόνο 2,5 δισεκατομμύρια ως στόχο όταν μπορούμε κάλλιστα να αυξήσουμε το ποσοστό των καταναλωτών στην Ευρώπη. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Σας ευχαριστώ για την ε, δουλειά σας και την συνεισφορά σας ε, στην ευρωπαϊκή οικοδόμηση. Για τις κρατικές προμήθειες και δημοπρασίες το 12. Εμείς θα είμαστε από πίσω σας για τα θέματα αμοιβαιότητας ε, στην ε, σε, εμπορικές, ε, σε ευρωπαϊκές συναλλαγές. Ε, πήγατε στην Κίνα πρόσφατα και θέλω να ξέρω τι σας είπαν οι Κινέζοι για το άνοιγμα των δημοπρασιών εκεί. και για τις άμεσες επενδύσεις των ε, μη ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε ευρωπαϊκό έδαφος. Κύριε Επίτροπε, εγώ μιλώ εκ μέρους όλων των συναδέλφων, πιστεύω. Είδαμε αυτό το κείμενο, το μας παρουσιάσατε. Το θέμα είναι ότι εδώ θέλουμε ποιότητα. Ε, η ποιότητα είναι πάρα πολύ καλή, δεν λέω. Σε αυτό το προϊόν δεν έχω κανένα πρόβλημα με την ποιότητα αλλά ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες όταν έχουμε ένα αποσταγμένο προϊόν και το θεωρώ αυτό την ενιαία πράξη προϊόν απόσταξης και όταν δεν είναι καλό το προϊόν το αποσταγμένο παθαίνεις πονοκέφαλο Α, ο, ο κύριος και η κυρία Ράπτη. Κυρία Ράπτη τελευταία. Ε, λοιπόν, επειδή μιλήσαμε για προϊόν απόσταξης, θα σα πω ότι στην Ελλάδα και δει στην Κρήτη έχουμε το καλύτερο προϊόν απόσταξης, ρακή. Έτσι λοιπόν ο Επίτροπος ίσως χρειάζεται να δοκιμάσει και λίγη ρακή για να λειτουργήσει ακόμα καλύτερα. Ε, υπάρχουν τρεις μοχλοί Υπάρχουν τρεις μοχλοί στους οποίους θέλω να αναφερθώ ο δεύτερος, ο όγδος και ο δέκατος. Ε, στους, τρεις αυτούς, στους τρεις αυτούς μοχλούς ο κύριος Μπαρνιέ είναι ουσιαστικά α, συνυπεύθυνος. Νομίζω ότι ο μοχλός ο δέκατος που έχει να κάνει με την κοινωνική συνοχή είναι ο κυριότερος για να λειτουργήσουν και ο δεύτερος μοχλός που αφορά την κινητικότητα των εργαζομένων και ο όγδος μοχλός που αφορά την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Το ερώτημά μου είναι πότε προβλέπετε να καταθέσετε την πρότασή σας για την κοινωνική συνοχή. Um, I'm going to be very indulgent Θα είμαι πολύ επίκης, διότι έμεινε ένας ομιλητής, οπότε δίνω το λόγο στην σκιώδη συγγήτρια, που ήταν και πολύ δραστήρια. Χειροκροτώ το 4, 8, 9 και 12 από αυτές τις προτάσεις. Πολύ, πολύ επικοδομητικές. Μία ερώτηση επί του 10. Λέτε ότι θα προτείνετε νομοθεσία εφαρμόσιμη σε όλους τους τομείς η οποία θα βελτιώνει την ελευθερία της εγκατάστασης και θα προωθεί τα σεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα. Του τέστην. Σας ευχαριστώ όλους ε, για την, τον δυναμισμό σας ε, στις ερωτήσεις αυτές. Θα απαντήσει ο Επίτροπος και θα καταβάλει κάθε προσπάθεια. Κάποιο μικρόφωνο ανοιχτό. Α, Συγγνώμη για αυτέ τι τόσο τηλεγραφικέ απαντήσει. Σα ευχαριστώ για την εκτίμησή σα, ε, κυρία μου. Τώρα, και αυτό που είπε η κυρία Ράπτη ως πολύ σημαντικό θέμα, δηλαδή την κοινωνική συνοχή, σας λέω ότι πρόκειται για ένας από τους όρους ε, για να πετύχουμε μια υφόρο λύση με ολοκληρωμένη αγορά και καινοτομία τα πράγματα συμβαδίζουν με την κοινωνική συνοχή. Και στην εισαγωγή εμείς αναφέρουμε τη δέσμευση της Κομισιόν υπό το πνεύμα που κάναμε για την οδηγία, με την οδηγία για τις υπηρεσίες από κοινού με σας και διευκρινίζουμε ότι, ότι ξέρω ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει συμβατότητα της εσωτερικής αγοράς με την ποιότητα, την πρόσβαση της ποιότητας ε, ε, στις καθολικές υπηρεσίες, υπηρεσίες καθολικού γενικού συμφέροντος. Κύριε Βάντερ, ε, λοιπόν, όταν μου λέτε τι, τι κάνουμε για τους πολίτες, μας είστε εκπρόσωπος των πολιτών. Και εγώ δεν είμαι πια ένας υπερτεχνοκράτης. Και εγώ βουλευτής ήμουν σαν και εσάς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν είμαι ένας υπερτεχνοκράτης βρυξελιώτης, είμαι ένας πολιτικός. Κυρίες και κύριοι, έχουμε με ζωτική σημασία δουλειά να κάνουμε. Βρισκόμαστε σε, μια, σε ένα σταυρικό σημείο ή σε κάθε χώρα θα την κερδίζει ο λαϊκισμός στην υπόθεση, τη δική σας ή τη δική μου, και με τον λαϊκισμό μετά θα έρθει ο προστατευτισμός και βλέπουμε την πρόθεση παντού και τέρμα εσωτερική αγορά. Και τέρμα και το ευρωπαϊκό σχέδιο. Αυτό σας λέω. Ή θα σταθούμε ικανοί, είτε είμαστε αριστεροί είτε δεξί. Διότι ξέρετε το ευρωπαϊκό σχέδιο δεν είναι αριστερό ή δεξιό, μας ανοίξει σε όλους. Λοιπόν, ή θα αποδείξουμε ότι θα πρέπει να εξηγήσουμε πώς δουλεύει το σύστημα. Όλοι μας θα το κάνουμε και όλοι πρέπει να το μάθουμε πώς δουλεύει. Δεν υπάρχουν χιλιάδες απαντήσεις για το πώς κερδίζεται αυτή η δημοκρατική πρόκληση. Υπάρχει ένα τεράστιο πολιτικό ζήτημα, μια πολιτική κρίση μαζί με την οικονομική κρίση. Κύριε Μπουσουτήλε, για τη δυνατότητα των ΜΜΕ να βγούνε από την περιφέρειά τους και από τα σύνορά τους. Μα φυσικά υπάρχει το ηλεκτρονικό εμπόριο που πρέπει να διευκολύνουμε και θα σας παρουσιάσω τον αναθεωρημένο πακέτο, καλύτερα μια ανακοίνωση για το ηλεκτρονικό εμπόριο σχετικά με τις ε, εξαγωγές, οι δυνατότητες της, στην πρόσβαση των επιχειρήσεων στις δημοπρασίες, η ηλεκτρονική υπογραφή, η ηλεκτρονική ταυτότητα, στο ίντερνετ, ε, τα συστήματα μετάφρασης για τις γλώσσες, για τις ΜΜΕ, αυτό που κάναμε δηλαδή για τις ΜΜΕ είναι πάρα πολύ Αυτό για να διευκολύνουμε δηλαδή την κατάσταση. Κύριε Βέιλερ, Ξέρω ότι πολλές φορές ο δημοκρατικός χρόνος ξεπερνάει τα όρια της υπομονής. Αλλά κι εσείς εδώ χρειάζεστε ε, το χρόνο για να σεβαστείτε τα κείμενα και όλα τα σχετικά. Για τις οικονομικές υπηρεσίες, αυτό το οποίο προχωράει πιο γρήγορα είναι οι χρηματοπιστωτικές αγορές από τις δημοκρατικές διαδικασίες. Αλλά και εμείς κάναμε ό,τι μπορέσαμε, όπως είπε και ο Πρόεδρος μας, 14 μήνες είμαι επίτροπος. Η έκθεση Μόντι ξεκίνησε πριν. Ολοκληρώθηκε στην άνοιξη του 2010 και πριν ολοκληρωθεί το πόρισμα της έκθεσης Μόντι ξεκίνησα μαζί, μπήκα, στρωθήκαμε στη δουλειά μαζί τον πρόεδρο Μπαρός, εγώ και άλλοι 12 συνάδελφοι και είχαμε και την ε, ε, τις ακροάσεις αυτούς τους μήνες και καταλήξαμε. Απάντησα και στον κύριο Αρίας που τον ευχαριστώ για το ηλεκτρονικό εμπόριο και για την ανακοίνωση που θα παρουσιάσω σε μερικούς μήνες. Κύριε Ρίπ, πήγα στην Κίνα για να μιλήσω για τις ε, ε δημόσιες αγορές, για τις δημοπρασίες. Ε, μιλήσαμε για την αμοιβαιότητα, μιλήσαμε για τα θέματα για τα οποία δεν υπάρχει αμοιβαιότητα στην Κίνα. Δεν μπορούν οι επιχειρήσεις μας να παρέμβουν σε πάνω από το 23% του κεφαλαίου των επιχειρη... κινέζικων επιχειρήσεων. Οι ασφαλιστικές μας εταιρείες δεν μπορούν να υποβάλουν ε, προσφορές για τις ασφάλειες ζωής ή για την ασφάλιση αυτοκινήτων ή για την ασφάλιση μετοχών στην Κίνα. Βέβαια δεν μου δώσαν αρνητικές απαντήσεις. Ο διάλογος συνεχίζεται. Όπως επίσης και με τα θέματα των, της διαφάνειας, των μέσων διαφάνειας για να δούμε ποιος αγοράζει τι στην Ευρώπη. Ε, με βοσθητοποίησε η πρόταση της κυρίας Ράπτη να πίνω αρκετό ρακί για να κρατάω τη φόρμα μου όχι βέβαια υπερβολικά, αλλά η κοινωνική συνοχή είναι κάτι το πολύ σημαντικό για την εσωτερική αγορά. Λοιπόν, αυτή αυτό το αυθόρμητο χειροκρότημα αξίζει πολλά. Σας ευχόμαστε ό,τι καλύτερο εκεί που πάτε, στη, ε, στην Ελβετία είπε, ο πρόεδρος στη Σουηδία πάει, ο επίτροπος στη Σουηδία διορθώνει, ο πρόεδρο. Λοιπόν, η κυρία Ρούλε και η κυρία Μανιουέλ θα πάρουν τη θέση, τη, την έδρα εδώ. Yes, I guess, I guess, I guess, I guess. Je Όποιος θέλει να βγει, να βγει στα γρήγορα σας παρακαλώ για να αρχίσουμε και πάλι τη δουλειά μας. Μέχρι τις 6.30 έχουμε πολύ σοβαρά ζητήματα τα οποία ε, αναφέρθηκαν και στη Single Market Act. Θα συνεχίσουμε λοιπόν στο θέμα του εξυγχρονισμού των κρατικών προμηθειών. Δίνω το λόγο στην εισηγήτρια την κυρία Χάιντε Ρούλε. Ευχαριστώ. Καταρχάς, να σας ε, πω το χρονοδιάγραμμα, τι τέλο πάντων έχει γίνει, τι τρέχει και να ενημερώσω τους συναδέλφους τι θα γίνει φέτος. Γίνεται η διαβούλευση με την Κομισιόν για το θέμα πράσινη βίβλος, κρατικές ε, προμήθειες. Μέχρι τις 17 Τετάρτου θα έχει ολοκληρωθεί. Ε, επίσης ε, έχουν ε, ανακοινωθεί διάφορες μελέτες, θα γίνει ένα συνέδριο στις 30 Ιουνίου όπου θα συζητηθούν οι επιπτώσεις της διαβούλευσης για την πράσινη βίβλο και επίσης θα συμπεράσματα από όλες αυτές τις μελέτες. Το δικό μας χρονοδιάγραμμα είναι πολύ καλό διότι πρέπει να συμπίπτει και με την Κομισιόν. Η έκθεσή μας θα συζητηθεί εδώ στην Επιτροπή 11-12 Ιουλίου, θα έχει και μεταφραστεί, προθεσμία τροπολογιών 19 Ιουλίου και ψηφοφορία σε εμά στην ΙΜΚΟ 19 Σεπτεμβρίου στην Ολομέλεια τη 2η του Οκτωβρίου. Άρα καλά τα πάμε, διότι μέχρι το τέλος του χρόνου έχει ανακοινώσει η Κομισιόν και την αναθεώρηση, οπότε οκτώβριο ταιριάζει πολύ καλά. Το μόνο που με στεναχωρεί είναι κανένας ε, δεν μιλάει στο, στην πράσινη βίβλο για τις ηλεκτρονικές προμήθειες, το e-procurement που συμπεριλαμβάνεται στη δική μου γνωμοδότηση. Έχουν ολοκληρωθεί διαβουλεύσεις και εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να συμπεριλευθεί αυτή η γνωμοδότηση και το θα το συζητήσουμε και στην ακρόασή μας στις 24 Μαΐου. Όχι και γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία η ανάπτυξη του συστήματος e-procurement, διότι έχουμε διάφορα ηλεκτρονικά συστήματα τα οποία θα συμβαδίσουν και πρέπει να είναι συμβατά το ένα με το άλλο, να λειτουργούν με open source ε, λογισμικό και γι' αυτό η ευρωπαϊκή, το ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να προτείνει ε, ε, κάτι σοβαρό. Εγώ πιστεύω ότι το e-procurement μπορεί να μπει άνετα ε, στην αναθεώρηση για τις κρατικές προμήθειες. Τώρα, επί της ε, ουσίας, ο στόχος της Κομισιόν ε, στην πράξη της εσωτερικής αγοράς είναι καταρχάς να γίνει ευρύτερη χρήση των κρατικών προμηθειών για την αηφόρο ανάπτυξη, τις καινοτομίες και τις πράξεις κοινωνικής, τα προγράμματα κοινωνικής ευθύνης. Όμως η οδηγία αυτή υποκρατικών προμηθειών έχει προβλήματα. Όταν μιλάει κανείς με τους ενδιαφερόμενους, διαπιστώνει την βαριά γραφειοκρατία, τις δύσκολες διαδικασίες. Άρα λοιπόν στην αναθεώρηση πρέπει, η δικιά μας τώρα, η επόμενη αναθεώρηση πρέπει να γίνει πολύ πιο καλά από το 2004. Ήδη έγινε προσπάθεια πλούστευσης ε, της ε, οδηγίας ανάθεσης ε, κρατικών προμηθειών ε, αλλά δεν ήταν επιτυχής. Το 2004 η οδηγία μεταφέρθηκε στο κρατικό, στα κρατικά δίκαια, αλλά τα προβλήματα εμφανίστηκαν και τελικά όλο το πλέγμα κρατικών ε, προμηθειών και αναθέσεων όχι μόνο δεν απλουστεύθηκε, έγινε πιο περίπλοκο και πιο ακριβό. Το ερώτημα λοιπόν τώρα είναι τι λύσεις προτείνουμε, πώς μπορούμε να φροντίσουμε αυτή τη φορά η αναθεώρηση να επιτύχει. Καταρχάς πρέπει το νομοθετικό πλαίσιο να είναι πιο, ε, ε, πιο ευκρινές, να διευκρινιστούν πιο σαφές. Εάν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε περισσότερο το πλέγμα των κρατικών προμηθειών για τους πολιτικούς μας στόχους, πρέπει να χρησιμοποιούνται οι κρατικές προμήθειες και όλες αυτές οι διατάξεις και για την αηφορία και για τις καινοτομίες. Άρα δεν πρέπει να στοχεύουμε συνέχεια ε, στην ε, φθηνότερη προσφορά ενός μειοδοτικού διαγωνισμού ας πούμε, όπως γίνεται συνήθως, Ιδιαίτερα όταν οι, οι κρατικές αρχές ε, δεν, δεν ήξεραν ακριβώς τι διατάξεις ισχύουν και ιδιαίτερα στις κοινωνικές υπηρεσίες όπου είναι δύσκολη η σύγκριση τιμών, πολλές φορές για λόγους ευκολίες κατέφευγαν στη φτηνότερη λύση η οποία δεν ήταν ούτε πολύ αηφόρος ούτε πολύ καινοτομική. Ε, έχω πολλά παραδείγματα από την Ολλανδία. Θα σας το διαβάσω για να σας εξηγήσω το επιχείρημά μου. Μία ε, μία επαρχία της Ολλανδίας ήθελε να αγοράσει πρίντερες, εκτυπωτές, υβριδικούς εκτυπωτές και πίστευαν ότι αυτές, ε, αυτοί οι εκτυπωτές νέες τεχνολογίες προσφέρουν ε, χίπλων εκτήματα. Δεν ήταν εύκολη η σύγκριση με τους παλαιότερους εκτυπωτές και όλα τα πλεονεκτήματα δεν μπορούσαν να παρουσιαστούν εύκολα με, εκτός από ένα πλεονέκτημα και τελικά επιλέχθηκε η παραδοσιακά φτηνότερη λύση. Αυτό έγινε δυστυχώς διότι ήταν πολύ δύσκολη η συγκριτική πίνακες τιμών, ήταν δύσκολες οι συγκρίσεις εκτιμάτων και προδιαγραφών και κατέληξαν στο φτηνότερο. Ήδη από πέρσι είχα πει ότι θα πρέπει τα κριτήρια και τα, οι πίνακες σύγκρισης να είναι ενιαίοι αυτό το ερώτημά μας, ε, το αίτημά μας δεν απαντάται στο πράσι, στην πράσινη βίβλο. Τώρα η μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου είναι ένα βήμα, όμως αυτή η μεταρρύθμιση πρέπει να συνοδεύεται με συμπληρωματικές ε, δράσεις, όπως π.χ. να ξέρουμε το κόστος ανάλογα με τον κύκλο ζωής Πρέπει δηλαδή να μπορώ να συγκρίνω το κόστος ανάλογα με το life cycle, ανάλογα με τον κύκλο ζωής του προϊόντος, του έργου κλπ. Επίσης, είναι σημαντικό να μπορέσει η ευρωπαϊκή πλευρά να βοηθήσει την, επιλογή των κριτηρίων, ιδίω των κοινωνικών. Πολλές φορές ορισμένα προϊόντα που υπάρχει μια λυσίδα προμήθειας, χάνονται τα ίχνη των διαφόρων κόμβων προμηθειών και δεν είναι δυνατό να συγκρίνουμε πάντοτε τα προϊόντα τα οποία έχουν δικό του σύστημα πιστοποίησης και γι' αυτό πρέπει να βοηθήσει περισσότερο το ευρωπαϊκό επίπεδο. Μπορούμε να λέμε πολύ ωραία ότι οι κρατικέ αναθέσεις πρέπει να γίνονται με κοινωνικά κριτήρια. Όμως, αν δεν υπάρχουν και τα διαθέσιμα μέσα, τα διαθέσιμα εργαλεία για να κρίνουμε ποια είναι κοινωνικά ή όχι, δεν θα επιτύχουμε. Επίσης, είναι σημαντικό οι οδηγίες κρατικών προμηθειών να ε, στοχεύουν βασικά στις προμήθειες και να μην ασχολούνται με άλλα άσχετα ζητήματα. Μην χρησιμοποιούνται δηλαδή οι άσχετες εφαρμογές, όπως παραδείγματο χάρη χωροταξικές. Εδώ μιλάμε για ε, procurement, προμήθεια. Ε, επίσης είναι σημαντικό όλα τα, ερωτή, τα ζητήματα τα οποία έχουν σχέση με εσωτερικές διοικητικές διαδικασίες να μην επηρεάζονται από μη, μη εξωτερικές λειτουργίες. Δηλαδή να μην συγκρίνονται οι κρατικές ε, προμήθειες και οι κρατικές διαδικασίες ε, μονίμως με τις μη κρατικές. Ταυτόχρονα να χρησιμοποιούνται σύγχρονες μέθοδοι στην ανάθεση, όπως είπα, καινοτομίες, Επίσης, ε, σύγχρονες μέθοδοι διακήρυξης, διαβούλευσης, εξέτασης, εξελόγησης, όλα αυτά να είναι σύγχρονα μέσα. Και στην ακρόαση που θα κάνουμε, να τονίσω ότι αυτές οι μέθοδοι να παρουσιαστούν σύντομα σε εμά και να τις συζητήσουμε. Έχουν συμφωνήσει και οι σκιώδεις εισηγητές. Οι Σουηδοί ε, δίνουν το βάρος καταρχάς στην ποιότητα. Δηλαδή ζητούν σταθερές τιμές, αλλά η προκήρυξη του μειοδοτικού διαγωνισμού γίνεται βασικά με το κριτήριο της ποιότητας. Ωραία, καλέ είναι. Καλά είναι το κριτήριο των τιμών, αλλά πρωταρχικό ζήτημα είναι ποιότητα. Αυτά στη Σουηδία. Και εν συνεχεία με την διαφανή διαδικασία οι πολίτες μπορούν να παρακολουθήσουν την εξέλιξη της, ε, της διαδικασίας. Τα, βεβαίως και απλούστευση των διαδικασιών από την πλευρά των προμηθευτών, ιδίως όταν είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δηλαδή προεπιλεξιμότητα ε, να δούμε ε, εάν οι, μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι επιλέξιμες, εάν λειτουργεί σωστά η επιχείρηση, αν έχουν όλες τις διαδικασίες ε, λειτουργία που απαιτούνται για την απάντηση, για την εκτέλεση των υποχρεώσεών τους σε ένα διαγωνισμό κλπ. Αυτά είναι τα κεντρικά σημεία της γνωμοδότησής μου και μπορούμε να δείξουμε ότι και οι δύο πλευρές και για τον κρατικό τομέα αλλά και για τους προμηθευτές θα λειτουργήσει ένα σύστημα πιο απλό μέσα σε ένα ε, δομημένο νομοθετικό πλαίσιο έτσι ώστε εν τέλει θα μειωθεί ο ρυθμός των παραπώνων και των προσκομμάτων που παρουσιάζονται σήμερα. Μαζί με την αμοιβαία αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων, αυτή η διαδικασία κρατικών προμηθειών είναι πιο επιβαρημένη με παράπονα, με παραβιάσεις και με εμπόδια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την ποιότητα αυτής της παρουσίασης ενός κειμένου αρκετά δυσανάγνωστου και σύνθετου. Τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Σβάμπ. Ευχαριστώ. Η κυρία Ρούλε έδειξε τα κύρια σημεία της πράσινης βίβλου. Εγώ θα έλεγα για το ΕΛΚ, όπου δυστυχώ ο Φρανκ Έγκελ, που είναι σκιώδης ηγητής δεν μπορεί να είναι εδώ. Εμεί επιδιώκουμε βελτίωση της υπάρχουσας, των υπαρχουσών οδηγιών, αλλά όχι ακύρωση και στρέβλωση. Βεβαίως βελτιώσεις μπορεί να γίνουν σε πολλά σημεία, αλλά πρέπει να σκεφτούμε πολύ προσεκτικά αν αυτέ οι ιδέες θα οδηγήσουν στο στόχο μας. Δηλαδή ο στόχος μας είναι να υλοποιήσουμε τις υποσχέσεις μας. Ε, ομολογώ ότι εξεπλάγει όταν ένας από αυτούς τους μοχλούς στην ενιαία πράξη είναι η αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου των διαδικασιών ανάθεσης κρατικών προμηθειών. Εμείς έχουμε μια οδηγία από το 2004 που ενδέχεται να μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω. Αλλά όπως είπε και η Κομισιόν, στο θέμα των παραχωρήσεων δεν έχουμε τίποτα. Τώρα δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει τόσο πολύ να προωθήσουμε το θέμα αυτής της οδηγίας. Βεβαίως είπα ότι υπάρχουν ε, δυνατότητες βελτίωσης και από τις δύο πλευρές, και προμηθευτές και, και κρατικές υπηρεσίε. Δεν ξέρω βέβαια αν το κρατικό πλαίσιο αυτό λειτουργεί σωστά. Πολλές φορές δημιουργούνται ε, υπερβολικά αυστηρές εφαρμογές μιας νομοθεσίας για περιορισμό του μηχανισμού ανάθεσης και προκήρυξης όσον αφορά το διάλογο για την ανταγωνιστικότητα, διαπιστώσαμε πολύ ε, σωστά ότι σε μία σειρά ε, κρατών μελών δεν εφαρμόζεται η οδηγία. Ε, πρέπει να δούμε πριν προχωρήσουμε να κάνουμε μία αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης. Πώς έχει μεταφερθεί στο δίκαιο ή δεν έχει μεταφερθεί και πώς εφαρμόζεται η οδηγία. Οι οδηγίες. Ακούσαμε το Ολλανδικό παράδειγμα. Εγώ έχω ένα άλλο παράδειγμα. Ένας που κατασκευάζει εξιονιστικά μηχανήματα για την τοπική αυτοδιοίκηση. Ο οποίος για κάθε μηχάνημα, επειδή κάθε, κάθε κράτος μέλος έχει διαφορετικές προδιαγραφές για τα εκχιονιστικά μηχανήματα, χρειάζεται ο κατασκευαστής να φτιάξει διαφορετικά μηχανήματα ή διαφορετικά εξαρτήματα, εν πάση περιπτώσει κινητήρες, στους εκχιονιστήρες του. Ένα προσπαθεί λοιπόν να φτιάξει μηχανήματα τα οποία είναι φιλικά στο περιβάλλον, επιβαρύνεται τόσο πολύ και επιβαρύνεται και ο φορολογούμενος εν τέλει με όλη αυτή την περιπλοκότητα των προδιαγραφών και των διατάξεων. Το θέμα είναι και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπορούν να κάνουν τις προσφορές τους ε, ε, με απλό τρόπο και σαφή ε, και ο κρατικός μηχανισμός από την άλλη πλευρά να είναι ξεκάθαρο στο τι ζητάει. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει οπωσδήποτε να ασχηθούν έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις προσφορές, στους ομοιοδοτικούς αυτούς διαγωνισμούς. Τι μπορούμε λοιπόν να βελτιώσουμε. Αυτό πρέπει να κοιτάξουμε. Όχι μόνο νομοθετικά, αλλά και στην πλευρά της εφαρμογής. Σίγουρα η εφαρμοστική πλευρά έχει δυνατότητες βελτιώσεων. Ευχαριστώ. Ε, ζητώ συγγνώμη, αλλάξαμε θέσεις. Λοιπόν, Είμαι σκιώδης ε, στο θέμα αυτό και με τη Χάιντι συμφωνώ σε πολλά. Είναι βασικό να γίνει η αναθεώρηση της νομοθεσίας των κρατικών προμηθειών στην Ευρώπη. Το λέμε γιατί κανονικά ε, πρέπει να υπάρξει μια, νέα στρατηγική, ε, μια καλή στρατηγική για μια νέα ανάπτυξη που ανταποκρίνεται σε κοινωνικά κριτήρια αλλά και σε περιβαλλοντικά. Για όλες τις κοινότητες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τις οποίες γίνεται μεγάλος λόγος στη Single Market Act, είναι σημαντικό η νομοθεσία να είναι ξεκάθαρη και απλούστερη. Εγώ θα δώσω ένα παράδειγμα γιατί ε, στο χώρο που ζω, στην κοινότητα που ζω, ε, υπάρχει ε, ε, η δυνατότητα να γίνει μια ομαδική αγορά βιβλίων για τις βιβλιοθήκες και τα σχολεία. Το γεγονός ότι έχει επιλεγεί μια τοπική επιχείρηση, η οποία ήταν ελάχιστα ακριβότερη από ότι μια παρισινή επιχείρηση, απλώς και μόνο επειδή θέλαμε να διατηρηθούν θέσεις εργασίας τόπου Και όταν έγινε ε, η σούμα του κόστους αγορά και του οικολογικού κόστους της μεταφοράς, εμείς ε, ως κοινότητα επιλέξαμε αυτή την ε, επιχείρηση. Χρειάζεται όμως να δικαιολογούμαστε μόνο και μόνο επειδή δεν αγοράσαμε ε, μόνο το, το ε, Δεν ήταν δηλαδή μέχρι τώρα κριτήριο η ποιότητα. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις επίσης. Τώρα, το δίκαιο εμπόριο πραγματικά αποτελεί ένα όραμα αλληλεγγύης που ε, μπορεί να προσφέρει σε ολόκληρο τον κόσμο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλήσαμε για την παγκοσμιοποίηση, για ολόκληρο τον κόσμο. Η Ευρώπη παίζει ρόλο ε, αλλά να παίζει ρόλο και ως υπόδειγμα, ως παράδειγμα στο δίκαιο εμπόριο ε, δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψη στις κρατικές προμήθειες. Αυτό αναφέρθηκε και στο Single Market Act ε, του Επιτρόπου Μπαρνιά. Η αμοιβαιότητα στους κανόνες των κρατικών προμηθειών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης, βιομηχανικών χωρών και αναδειωμένων χωρών. Αυτό το θεωρώ σημαντικό και για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπήρχε ως κριτήριο μέχρι τώρα. Όταν μιλάμε επίσης για ποιότητα, υπάρχει η ποιότητα των δικαιωμάτων των εργαζομένων αλλά και των προϊόντων και φυσικά είναι το θέμα της υπεργολαβίας. Οι μεγάλες κρατικές προμήθειες, οι κατασκευαστικές έχουν ένα θέμα ε, υπεργολαβίας γιατί μέχρι τώρα η νομοθεσία ήταν ανεπαρκέστατη. Και δεν συμφωνώ με τον κύριο Σβάμπ εδώ, γιατί εδώ έχουμε έναν λόγο να πούμε και δεν είναι θέμα μόνο να αποφασίσει η ευρωπαϊκή δικαιοσύνη. ευχαριστώ. Το πράσινο βιβλίο της Κομισιόν έχει πάρα πολύ καλές ιδέες και προτάσεις. Και γι' αυτό κυρία Ρούλε περιμένουμε με ανυπομονησία τι θα προκύψει από εσά. Ιδίως το θέμα που δεν υπάρχει στην πράσινη βίβλο, αλλά εσείς το θίξατε. Στην ηλεκτρονική ανάθεση, η ηλεκτρονική διαδικασία, το e-procurement. Ε, επίσης, είναι πολύ σημαντικό το κόστος ε, ανάλογα με τον κύκλο ζωής Ωραία είναι να δίνουμε το φτηνότερο, αλλά δεν έχει τη δυνατότητα να επιζήσει πολλά χρόνια ένα προϊόν ή ένα αγαθό. Λοιπόν, ε, χρειαζόμαστε και διαφορετικά κριτήρια, όχι μόνο το κόστος, τη τιμή. Γι' αυτό πιστεύω ότι το συνολικό κόστος διάρκειας ζωής είναι μια πολύ, ένας πολύ σημαντικός ε, μοχλός, ένα σημαντικό εργαλείο, το οποίο πρέπει να ληφθεί υπόψη στην όλη εξέταση της προσφοράς. Βεβαίως πρέπει να αυξήσουμε, να εξασφαλίσουμε τη διαφάνεια των διαδικασιών. Αλλά το είπατε και εσείς κυρία Ρούλε, είπατε ότι πάντοτε στην προκήρυξη λαμβάνονται υπόψη και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εμείς αυτές θέλουμε κατά προτεραιότητα να υποστηρίξουμε ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις προκηρύξεις χωρίς να επιβαρύνονται υπερβολικά με τη γραφειοκρατία. Δεν έχουν και τον καιρό ε, να διαθέσουν χρόνο να εξετάσουν όλο το, το, το, πλέγμα των γραφειοκρατικών διαδικασιών και γι' αυτό ακριβώς κερδίζουν συνεχώς οι μεγάλες επιχειρήσεις. Είναι λοιπόν στο συμφέρον και των δύο πλευρών η απλοποίηση των διαδικασιών, η βελτίωση της διαφάνειας και να δούμε τι θα γίνει με αυτή την ιδέα του κύκλου ζωής. Πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση διότι συνήθως εξετάζουμε το βραχυπρόθεσμο κόστος, πόσο κοστίζει σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Αλλά άμα εξετάσουμε τη μακροπρόθεσμη προοπτική, ε, αλλάζουν τα πράγματα. Ε, αυτό έχει συμβεί στο κρατήδιό μου, στο Ζάρλαντ. όταν ε, αναγκάστηκαν να εκτιμήσουν τις ζημιές ε, δεν μπόρεσαν να έχουν ακριβή στοιχεία διότι όλη η εκτίμηση το της προσφοράς είχε γίνει για, το βραχυπρό, για βραχυπρόθεσμη, για μικρή διάρκεια και όχι για την ε, μακροπρόθεσμη διάρκεια όπου θα μπορούσαν να είχαν συνυπολογίσει τα ελαττώματα, τις ζημίες κλπ. Για, αυτά έχω να πω προς το παρόν και γι' αυτό περιμένουμε να δούμε τι θα μας παρουσιάσετε επαναλαμβάνω, και στη διαδικασία προκήρυξης πρέπει ε, να επισέρχεται το στοιχείο της καινοτομίας. πολλές, ε, έχω πολλά παραδείγματα που δείχνουν ότι παραδείγματο χάρη στον κατασκευαστικό τομέα σπιτιών ε, έκαναν μια καινοτομική πρόταση και έτσι μπόρεσε και στην εφαρμογή ε, να βελτιωθεί το όλο πρόγραμμα. Λοιπόν, ευελιξία, καινοτομίες, αλλά όλα αυτά πρέπει να ε, καλύπτονται από ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, ένα δομημένο πλαίσιο μέσα στο οποίο θα ενταχθεί η διαδικασία προκήρυξης, ε, προσφοράς ε, και ανάθεσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κρότσμαν. Παίρνω τη σειρά μου ως σκιώδης της ομάδας μου. Ζητώ συγγνώμη στην κυρία Ρούλε που δεν παραβρέθηκα όταν εκείνη έκανε την παρουσίασή της. Έχουμε συνεργαστεί όμως στο προηγούμενο θέμα και συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό μαζί της. Κύριο Κρότσμαν και η κυρία Βενιού και αυτοί το είπαν κατά τον ίδιο τρόπο. Ότι δηλαδή πρέπει να επικεντρωθούμε στο τι θέλουμε από αυτό το σύστημα κρατικών προμηθειών. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι, και αν ρωτήσετε τους εμπλεκόμενους, αυτούς που χρησιμοποιούν το σύστημα, θα ακούσετε ότι η διαδικασία έχει ε, κυριαρχήσει στο αποτέλεσμα. Δηλαδή υπάρχει αυτό το πρόβλημα στις δημόσιες προμήθειες. Δεν ξέρω αν κάποιος άλλος εδώ ξέρει κάτι άλλο, μπορεί να μας το πει. Αλλά η κυρία Ρούλευ νομίζω ότι συμφωνεί μαζί μου. Αυτοί που ασχολούνται με τις κρατικές προμήθειες ασχολούνται περισσότερο με την τήρηση των κανονισμών παρά για να κάνουν καλές αγορές και να ασχοληθούν με την ποιότητα του αποτελέσματο. Και είμαστε ευαίσθητοι σε πολλά από τα θέματα που ήδη έχουμε συζητήσει για το γεγονός ότι θέλουμε περισσότερο περισσότερες μικρές επιχειρήσεις να εμπλακούν στις κρατικές προμήθειες γιατί παραδίδουν ενδιαφέροντα, ελκυστικά και καλά προϊόντα σε χαμηλότερο ε, κόστος και σε πολλές περιπτώσεις καλές θέσεις εργασίας. Άρα δεν είμαστε αλτρουιστές, δεν θέλουμε να συμμετέχουν μόνο και μόνο επειδή είναι μικρομεσαίες, αλλά επειδή θα κάνουν καλή δουλειά. Το σύστημα το ενθαρρύνει κάτι τέτοιο. Και το θέμα της, ε, ε, ε, καινοτομία. Ξέρετε ότι μένα με καίει αυτό, το υποστηρίζω και ε, πλέον ε, έχει, αναλάβει, έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις. Αν μια δημόσια αρχή επιθυμεί να καθορίσει μια πιθανή λύση με βάση το τελικό αποτέλεσμα και μετά πάει και ψάξει καινοτόμες επιχειρήσεις για να τις φτιάξουν αυτό το προϊόν και αυτό συμβαίνει σε κάποιες χώρες, τότε υπάρχουν τα εργαλεία να γίνει αυτό. Και πολύ σωστά μας ενδιαφέρει και το συνολικό κόστος ζωής της ποιότητας του αποτελέσματος, γιατί όλο και περισσότεροι οι άνθρωποι, περισσότεροι οι άνθρωποι θέλουν να επιλέξουν μια λύση με μικρότερο ε, ε, αποτύπωμα άνθρακα. Πώς θα μπορέσει να υπάρχει νομική ασφάλεια σε αυτό το θέμα. Υπάρχουν εταιρείε που μας παρακολουθούν και λένε ότι αυτό που θέλουμε είναι να δουλεύουν καλύτερα οι κανόνες, να είναι πιο ανταγωνιστική αγορά. Θα μπορέσουν οι ισχύοντες κανόνες να λειτουργήσουν ποτέ αποτελεσματικά. Αν δούμε τώρα τα αποτελέσματα σε σχέση με το πώς θα δοθεί μια όθηση στην ανταγωνιστική αγορά, η δική μου ο δικό μου Δήμο του Μπέρμιγχαμ, που είναι ο μεγαλύτερο του Ηνωμένου Βασιλείου, είναι μια πόλη περίπου ενό εκατομμυρίου. Ε, για να τηρήσει όλου του κανονισμού, κανονισμούς, έχει το μεγαλύτερο ε, προϋπολογισμό κρατικών προμηθειών του Ηνωμένου Βασιλείου και κάνει 200, 200 ε, δημοπρασίες, διαγωνισμούς εκτός Ηνωμένου Βασιλείου. Και άλλε εταιρείε το κάνουν αυτό, αλλά δεν αισθάνονται ότι τελικά η διαδικασία αποδίδει αυτό που θέλουν. Το γνωρίζει ο κ. Λάιν γιατί απαντώντας σε μια γραπτή ερώτηση ε, την περασμένη εβδομάδα, στο τέλος είπε ότι επιδιώκει ένα πιο ευέλικτο σύστημα που θα παρέχει αυτούς που ασχολούνται με τις κρατικές προμήθειες τα σωστά εργαλεία για να κάνουν αυτό που θέλουν να κάνουν και ένα σύστημα που θα είναι πολύ λιγότερο γραφειοκρατικό, λιγότερο σύνθετο, λιγότερο δαπανηρό και αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ επιδιώκω μια ριζική μεταρρύθμιση του συστήματος. Δεν μ' αρέσει το ε, ισχύον καθεστώς που λέει ότι ό,τι την αλλάξει είναι καλό. Δεν το πιστεύω αυτό και πιστεύω ότι και εσείς δεν το πιστεύετε. Θεωρώ ότι ο τρόπος που έχει διατυπωθεί η πράσινη βίβλος και οι ε, ερωτήσεις έχουν διατυπωθεί θα, θα είναι κάτι στο οποίο θα ανταποκριθεί η Κομισιόν. Θα είναι εξίσου ριζοσπαστική η Κομισιόν. Πραγματικά δεν θα πρέπει να φοβόμαστε να αντιμετωπίσουμε κάποια από τα θέματα που χρονίζουν. Είναι ρεαλιστικό το κατόφλιο, μήπως είναι πολύ χαμηλό, μήπως χρειάζεται κάποια άλλη διαδικασία να το μελετήσουμε. Και τέλος πρέπει να δούμε τα θέματα που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διαχείριση των κρατικών προμηθειών σε διάφορες χώρες, στις βέλτιστε πρακτικέ. Σα είπα, ήμουνα στην Νορβηγία. Εκεί η Νορβηγία, η Φιλανδία και Ιδίω η Σουηδία έχουν οργανισμούς κρατικών προμηθειών που έχουν σχέση με τις αρχές ανταγωνισμού τους. Γιατί θεωρούν ότι αυτά τα δύο είναι απολύτως αλληλένδετα. Είναι κομμάτι της ανταγωνιστικής αγοράς να γίνει καλή η λειτουργία των κρατικών προμηθειών. Όμως σε μεγάλο βαθμό υπάρχει και η καινοτομία εδώ. Άρα στη Φιλανδία, Σουηδία και Νορβηγία ο κόσμος προωθεί την καινοτομία και υπάρχει ειδικό τμήμα που ασχολείται εκεί με τις κρατικές προμήθειες και προσπαθούν να ταιριάξουν τις απαιτήσει των κρατικών ε, προμηθειών με λύσεις που προέρχονται από πανεπιστήμια και άλλες σχολές. Εγώ θυμάμαι ότι 2004 στη διάρκεια της νομοθεσίας συμπεριλάβαμε μια αιτιολογική σκέψη που λέει ότι οι χώρες θα πρέπει να μελετήσουν τον τρόπο που λειτουργούν οι κρατικές προμηθειές και να το βελτιώσουν. Ξέρω ότι υπάρχουν διάφορα δίκτυα βέλτιστων πρακτικών, αλλά λειτουργούν όσο καλά θα έπρεπε. Τελικά νομίζω για μία ακόμα φορά, με βάση αυτά που είπε στην προηγούμενη έκθεσή της κυρία Ρούλε και με χαίρομαι που είχαμε τη Σοφία την, ως Επιτροπή να την συνεχίσουμε αυτή τη διαδικασία, ελπίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να διατυπώσουμε ε, ριζοσπαστικές ιδέες και να κάνουμε καλή συζήτηση από αυτών για να συμπληρώσουμε όλα τα στοιχεία που θα πάρει η Κομισιόν από τη δημοσίευση τη Πράσινη Βίβλου και πιστεύω ότι υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο μελετά κυρία Ρούλε για να μπορέσουμε να απορροφήσουμε κάποια από αυτά που θα υποθούν από τι μελέτε που θα προέρχονται τι μελέτε για να μπορέσουμε να συντάξουμε μία από τι σημαντικότερε εκθέσει μα σε αυτόν τον κύκλο του Κοινοβουλίου. Θεωρώ ότι ολοκληρώθηκε ένας, ο γύρος των σκιωδών. Ο κύριος Ντύρομι δεν είναι εδώ. Α πάρουμε τα μέλη της Επιτροπής, κυρία Βάιλερ και μετά κυρία Γκέπχαρτ και μετά όποιος άλλος θέλει να πάρει το λόγο. Κυρία Βάιλερ. Ευχαριστώ. Πραγματικά χαίρομαι που διαπιστώνω ε, μια γενική συμφωνία. Υπάρχουν διαφορετικές, λίγο διαφορετικές ε, ερμηνείες, αλλά γενικά με εκπλήτη συμφωνία. Πιστεύω ότι μετά τις επικρίσεις που κάναμε πριν από 6-7 χρόνια προσεγγίζεται περισσότερο την άποψή μας να ανυψώσουμε τα κατόφλια. Εάν οι τιμές κατοφλίου αυξηθούν, σηκωθούν, ε, αυξηθούν, τότε ε, ε, αυτό θα γίνει στο σπίτι του καθενός, δεν θα γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δηλαδή στα κράτη-μέλη, ε, και σύμφωνα με τον καλύτερο τρόπο που επισημεί ο, καθέ, ο Εγώ πιστεύω ότι όλη αυτή η εργασία στο ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να έχει ένα θετικό αποτέλεσμα και στα εσωτερικά της κάθε χώρας. Δηλαδή να αναθεωρήσει, να εξετάσει και να αξιολογήσει πώς λειτουργεί τέλο πάντων όλη η διαδικασία κρατικών προμησιών. Πολλές επικρίσεις είχαν ακουθεί στο παρελθόν. Εγώ πιστεύω ότι το επίπεδο της απλούστευσης ε, όμως ε, πρέπει να είναι ευρωπαϊκό. Εμείς πάντοτε υποστηρίζαμε τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και βεβαίως και κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια τα, τα έχουμε υποστηρίξει και τα υποστηρίζουμε στεναρά συνέχεια. Ποτέ δεν υποστηρίζαμε εμεί τον ευθυνότερο μειοδότη. Υποστηρίζαμε το βέλτιστο, τον καλύτερο, λαμβάνοντα υπόψη αυτά τα κριτήρια. Και όταν ε, οι δήμαρχοι ή οι αντιδήμαρχοι είναι αρκετά ξύπνοι και ρωτούν τους πολίτες τους ποιο προτιμάτε αυτό το πρόγραμμα Α το οποίο είναι πιο καινοτομικό, πιο φιλικό στο περιβάλλον και έχει μεγαλύτερο κύκλο ζωής ή το Β, το οποίο είναι κατά δύο δεκάρες λιγότερο, ε, Οι περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν συμμετέχουν σε πανευρωπαϊκές προσφορές. Ε, είναι πολύ μεγάλα τα μεγέθη για τις μικρομεσαίες όταν είχαμε κάνει τις συζητήσεις ε, για το PPP, Private ε, Public Procurement, δηλαδή ε, συμμετοχή δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, είχαμε πει ότι πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα και στις μικρομεσές να συμμετάσχουν. Αυτή τη στιγμή δεν γίνεται όμως δυστυχώς. Στο μόνο σημείο που παρεμβαίνουν οι μικρομεσές είναι όταν υπεργολαβικά ας πούμε προμηθεύουν ορισμένα παραπροϊόντα στους μεγάλους προμηθευτές που εν συνεχεία λαμβάνουν τους, ε, την ανάθεση. Εγώ δεν ε, ε, πιστεύω ότι θα πρέπει να συμπεριληφθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ενισχυθούν όχι μόνο υπεργολαβικά, αλλά να μπορούν να συμμετέχουν ως ε, μειοδότε, ως, ως υποψήφιοι προς ανάθεση δηλαδή, χωρίς πάντοτε το μειοδοτικό στοιχείο του κόστους. Ευχαριστώ κυρία Βάιλερ, η κυρία Γκέπαρτ. Ευχαριστώ. Συμφωνώ και εγώ με αυτά που είπε η κυρία Βάιλερ. Πρέπει να πω ότι και εγώ εξεπλάγει θετικά με το επίπεδο της ε, σύμπτωσης απόψεων. Ε, είχα παρακολουθήσει στενά τις συζητήσεις στο παρελθόν για τις προμήθειες και είχαμε πει τα ίδια, ο φθηνότερος ή ο καλύτερος. Αυτό ήταν το πιο επίμαχο σημείο τότε στις συζητήσεις που έγιναν στην Επιτροπή. Και με πολύ στενή πλειοψηφία είχαν αποφασίσει τον βέλτιστο, τον καλύτερο. Σήμερα πραγματικά ε, ε, βλέπω ότι υπάρχουν και άλλες ε, γνώμες, άλλες απόψεις που ενισχύουν την πλειοψηφία για την επιλογή του καλύτερου. Πρέπει να δούμε ποια κριτήρια ποιοτικά μπορούν να εφαρμοστούν και πώς. Είναι αυτή η ποιοτική διάσταση τώρα την οποία διαπιστώνω και η οποία με χαροποιεί ιδιαίτερα η δεύτερη πτυχή όπου εν μέρη υπήρχε σύμπτωση απόψεων και πλειοψηφία ήταν οι τιμές κατοφλίων. Είχα τότε λάβει στοιχεία από γερμανικής πλευράς. Τους είχα ρωτήσει πόσες προκηρύξεις υπάρχουν, πόσες προσφορές εκτός Γερμανίας, τουλάχιστον στο, Γερμα... στο κρατήδιο της Βάρης ε, ε, Βάδης Βιρτεμβέργης και οι μη ε, τοπικοί ε, ήταν πάρα πολύ λίγοι. Πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε πού, σε ποιο επίπεδο πρέπει να θέσουμε το σωστό το κατόφλι, διότι δεν έχει κανένα νόημα να γίνονται προκηρύξεις σε τομείς όπου δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι και δεν ε, υποβάλλουν προσφορές. Άρα λοιπόν, όπου τα κατόφλια είναι κατάλληλα και όπου οι γραφειοκρατικές διαδικασίες μπορούν να απλουστευτούν, οπωσδήποτε πρέπει να το κάνουμε. Απλούστευση και βελτίωση. Το τρίτο ζήτημα όπου πιστεύω θα υπάρχει διάσταση απόψεων είναι ένα ερώτημα που με απασχολεί και δεν έχω απάντηση ακόμα. Αυτά τα κριτήρια της αηφορίας, κοινωνική διάσταση, όλα αυτά τα κριτήρια που θέλουμε να συμπεριλάβουμε. Θέλουμε να τα συμπεριλάβουμε στις ισχύουσες οδηγίες ως προαιρετικά ή ως υποχρεωτικά. Να είναι προαιρετικά κριτήρια ή υποχρεωτικά. Αυτό είναι το ερώτημά μου το οποίο θέτω. Δεν ε, έχω εγώ απάντηση, αλλά τουλάχιστον να τη σκεφτούμε. Να σκεφτούμε την απάντηση. Ευχαριστώ πολύ Άλλος κανείς. Α, η κυρία Σμιτ ήρθε από την ε, Κομισιόν. Θέλουμε να ακούσουμε τι έχετε να πείτε σε αυτά που ακούστηκε και μετά θα δώσω πάλι το ρόγο στην κυρία Ρούλιο και Σμιτ. Κυρία Σμιτ, καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ καταρχήν για το μεγάλο ενδιαφέρον που δείχνετε σε αυτή την, για αυτή τη μεταρρύθμιση. Είμαι ιδιαίτερο ευτυχή. Πραγματικά δικαιωνόμαστε στην άποψη ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το έργο και πραγματικά χαιρόμαστε που υπάρχει σύμπτωση απόψε ότι χρειάζεται μεταρρύθμιση γιατί ένα παράδειγμα. Η διαδικασία διαπραγμάτευσης σήμερα, σήμερα δεν επιτρέπεται όπως έχει σήμερα η οδηγία. Πρέπει λοιπόν να αλλάξει αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχουν πολλά που μπορούν να γίνουν σε δικό μας επίπεδο, αλλά και πολλά πρέπει να γίνουν σε επίπεδο κρατών μελών. Λοιπόν, θα επιστρέψω με όλες τις καινούργιες ιδέες που άκουσα σήμερα από την, στη Γενική Διεύθυνση Μάρκτ. Σαφώς είμαστε σε φάση προετοιμασίας, δεν θα επισέλθω στις λεπτομέρειες του περιεχομένου, όμως σαφώς συμφωνούμε με τα διάφορα θέματα που τέθηκαν ως σημαντικά, γραφειοκρατία, καλύτερη χρήση δημοσίων προμηθειών, βελτίωση των κοινωνικών, ε, της ε, κοινωνικής διάστασης και της καινοτομία, πολύ σημαντικό, ότι η έμφαση πρέπει να δοθεί στην ποιότητα. Πώς θα γίνει αυτό χωρίς να μπουν επιπλέον ε, γραφειοκρατικά εμπόδια στις συμβαλόμενες αρχές δεν είναι πολύ εύκολο. Το να φτιάξουμε κριτήρια ποιότητας για την καινοτομία και να πλουστεύσουμε ταυτόχρονα τους κανονισμούς. Θα είναι λίγο τετραγωνισμός του κύκλου, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε και ελπίζω θα καταλήξουμε με χρήσιμο τρόπο. Δύο λόγια για τη μεθοδολογία. Συμφωνούμε, είναι σημαντικό να υπάρχει διαφανής και ξεκάθαρη μεθοδολογία πριν επιβληθούν οι νέοι αυτοί κανόνες στους επιχειρηματίες. Προσπαθώ να είμαι σύντομη. Ένα πραγματάκι ακόμα για το διαμεθοριακό. Ξέρουμε ότι είναι χαμηλό το επίπεδο του διαμεθοριακού εμπορίου. Η κυρία Γκέπχαρτ ε, ρώτησε. Ε, το αξιολογούμε. Έχουμε το πλαίσιο της ισχύουσας οδηγίας. Η Κομισιόν το μελετάει. Θα σας το παρουσιάσουμε στη διάσκεψη του Ιουνίου που σας καλώ όλους Μέχρι εδώ. Ε, εκτός και αν έχετε κάτι το πολύ συγκεκριμένο με ρωτήσετε. Mm. Μπορείτε να μας πείτε πότε περιμέν, αναμένετε να δημοσιευθεί η περίληψη των απαντήσεων στη διαβούλευση της Πράσινης Βίβλου, γιατί αυτό είναι σημαντικό για το χρονοδιαγραμμά μας. Δουλεύουμε εντατικότατα. Δεν θα πάρει κανείς διακοπές. Δεν θα πάει κανείς διακοπές. Προσπαθούμε να το προετοιμάσουμε, να το έχουμε έτοιμο πριν την διάσκεψη. Αρχές Ιουνίου, αλλά δεν δεσμεύομαι. Επειδή όπως ακούστε την κυρία Ρούλε, θα κάνουμε και εμείς μια κρόση. Uh, κυρία Ρούλε, θέλετε να ανακεφαλαιώσετε. Έχετε χρονοδιάγραμμα, τι θέλετε. Okay. Σας εξήγησα το χρονοδιάγραμμα στην αρχή. Βάσει των μερομηνιών που έχουμε από την Κομισιόν. 12 Ιουνίου έχω. Καλά, μπορώ να συμπεριλάβω και τις προτάσεις της Κομισιόν εφόσον υπάρχει προθεσμία τροπολογιών, εντάξει. Άρα λοιπόν το χρονοδιάγραμμα συμπίπτει, είναι εντάξει, απλώς επιβεβαιώνω αυτά τα οποία είπε η Κομισιόν και από εσά, κύριε Πρόεδρε. Ε, πιστεύω ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο χρειάζεται οπωσδήποτε αυτή η αναθεώρηση, δεν είναι, revision. Αυτή η αναθεώρηση. Αυτή τη στιγμή πρέπει να το κάνουμε σωστά. Πρέπει πραγματικά η αναθεώρηση να γίνει σωστή. Έχει οριμάσει ο χρόνος, έχουμε την οικονομική κρίση, πολλές προκηρύξεις ε, διαγωνισμών ε, είναι αδρανείς, δεν προχωρούν περαιτέρω λόγω της οικονομικής κρίσης και αυτό καθυστερεί τις πάρα πολλά έργα και πολλές διαδικασίες. και όπως είπε και ο, ο δήμαρχός μας ε, πρέπει να συνεχίσουμε να, εργαστού, να εργαζόμαστε παρόλο που υπάρχουν κενά και ελλείψεις αλλά ε, εφόσον υπάρχουν αυτά τα κενά και τις καλύψεις και τα λάθη που έχουν γίνει πρέπει να μάθουμε τα παθήματα μαθήματα και να κάνουμε μια καλή αναθεώρηση. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για αυτή την καλή εισαγωγή. Υπότιτλοι Έχετε ήδη αρχίσει μια συζήτηση, κυρία Ρούλε, βλέπω, αλλά ήταν πολύ έντονη και ενδιαφέρουσα εισαγωγή σε αυτή την πολύ σημαντική έκθεση. Είχαμε την ευκαιρία να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση ακριβώς μετά την πρόταση του κυρίου Μπαρνιέ. Ε, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Υπάρχουν γνωμοδοτήσεις από πολλές επιτροπές, ε, κυρία Ρούλε, δεν ξέρω πόσες, αλλά οπωσδήποτε θα πρέπει να κάνουμε με την πράξη νέα αγορά, δηλαδή όλο και περισσότεροι να ζητήσουμε να μας δώσουν γνωμοδοτήσει, γιατί πρέπει να συζητήσουμε συζητηθεί εκτεταμένα στο Κοινοβούλιο. Δεν ξέρω πώς το κάνουν αυτό. Η Επιτροπή Εμπορίου το κάνει αυτό, δεν ξέρω ποιος άλλος. Πολλές επιτροπές ε, υποβάλλουν γνωμοδοτήσεις. Είχα στον κατάλογό μου και θα σας, το, θα σας τις πω γιατί πρέπει να συνεργαστούμε. Ήτρε, Ίντερ, απασχόληση, ένβη, νομίζω και η Ρέγγι δεν λέει, αλλά έχει, κάτι έχει κάνει η Περιφερειακή Επιτροπή και ελέγχου προπολογισμού. Επίσης, στην Επιτροπή των Περιφερειών υπάρχει θετική γνωμοδότηση. Πολύ ενδιαφέρουσα. Αναφέρεται στην ευελιξία, ε, στην τοπική αυτοδιοίκηση και η ΕΟΚΕ επίσης θα εκδώσει γνωμοδότηση. Μήπως θα πρέπει να τις καλέσουμε στην ακρόασή μας και όλες τις επιτροπές βεβαίως. Ναι, η Επιτροπή των Περιφερειών, βεβαίως. Και θα μιλήσω με τον πρόεδρο της Επιτροπής Μεταφορών, γιατί νομίζω ότι και εκεί κάτι πρέπει να γίνει. Τώρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, οπότε περνάμε στο επόμενο θέμα. Έχουμε... Είμαστε λίγο νωρίτερα. Περιμένουμε την κυρία εκπρόσωπο από την Κομισιόν. Έχει έρθει πολύ ωραία. Οπότε δεν ήθελα να ξεκινήσω πριν έρθετε εσείς. Χαίρομαι που βρίσκεστε εδώ. Όλη η ομάδα που δουλεύει είναι εδώ. κυρία Χάντσλικ είναι Welcome particularly, uh, who's worked with us before. Mrs. is... Κυρία Ρούλα, που δουλεύει πολύ σκληρά, είναι και πάλι ε, σκιώδης για τους πράσινους. Δεν ξέρω αν ο και εγώ θα συνεισφέρουμε σε αυτή τη συζήτηση διότι βλέπω ότι εκπροσωπείται το ECR. Λοιπόν, θα έχουμε γνωμοδότηση της Επιτροπής προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, που είναι η κύρια Επιτροπή, για την πρόταση για τον έλεγχο των ε, κινδύνων από σοβαρά ατυχήματα που συνεπάγεται ε, που εμπλέκουν επικίνδυνες ουσίες. Νομίζω όμως ότι αυτό έχει σχέση και με κάποια δική αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, κυρία Χάνσλικ, παρακαλώ να μας παρουσιάσει το θέμα και να μας πει ποια θα είναι η προσέγγισή της. Ε, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, πριν από λίγα λεπτά μόνο, στην Επιτροπή Περιβάλλοντος ολοκληρώθηκε ένα σεμινάριο για την τροποποίηση αυτής της οδηγίας. Μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, ένα ενδιαφέρον σεμινάριο με πολλές πληροφορίες και με αυτόν τον τρόπο είμαι ακόμα πιο... Έχω τη χαρά να σας μπορώ να σας δώσω περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό το θέμα που κατά την άποψή μου είναι θέμα που πρέπει να το αναλάβει η Επιτροπή μας στο πλαίσιο ε, της οδηγίας Σεβέζο 3. Λοιπόν, θα ήθελα να υπογραμμίσω αυτό που θίγει η οδηγία. Στόχος είναι να, η πρόληψη των σοβαρών προβλημάτων που έχουν σχέση με μεγάλες ποσότητες επικίνδυνων ουσιών ή μειγμάτων ουσιών και να περιοριστούν οι συνέπειες αυτών των προβλημάτων για τον άνθρωπο και για το περιβάλλον. Διότι αυτά τα σοβαρά ατυχήματα μπορούν να αποτελέσουν σοβαρή απειλή στους ανθρώπους, στην υγεία τους και στο περιβάλλον, όπως είπα τέτοιου είδους ατυχήματα μπορούν να αποβούν και πολύ δαπανηρά. Η οδηγία χωρίζει τους επιχειρηματίες που καλύπτονται από τις διατάξεις της, αυτούς που έχουν αυξημένο κίνδυνο και αυτούς που έχουν υψηλό κίνδυνο. Η βασική απέτηση της οδηγίας είναι να υποχρεωθούν οι επιχειρηματίες να καθορίσουν μια πολιτική πρόληψη σε περιπτώσεις σοβαρού ατυχήματο. Και σε υψηλού κινδύνου επιχειρηματίες υπάρχει η προϋπόθεση για εκθέσεις ασφαλείας και για την εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης ασφάλειας και προγράμματα, εσωτερικά προγράμματα ατυχημάτων. Η οδηγία περιλαμβάνει διατάξεις που αφορούν τις κρατικές αρχές, τις δημόσιες αρχές για εξωτερικά προγράμματα εκτάκτου ανάγκης, θέματα μέτρων ασφαλείας και για τους επιχειρηματίες υψηλού κινδύνου η, το φαινόμενο ντόμινο, το χωρο, η ταχύρητο χωροταξικός προγραμματισμός και οι επιθεωρήσεις. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 10.000 επιχειρηματίες οι οποίοι εμπλέκονται στις διατάξεις αυτής, το οποίο αφορούν οι διατάξεις αυτής της οδηγίας. Τώρα, στόχος αυτής της τροποποίησης της οδηγίας είναι η αλλαγή του συστήματος ταξινόμησης που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ε, ταξινόμηση των ουσιών. Θέλουμε δηλαδή να την ευθυγραμμίσουμε με το, τα όσα ισχύουν για την ταξινόμηση, την ε, ετικετοθεσία και τη συσκευασία διαφόρων μεικτών ουσιών. Καταρχήν το ένα καθορίζει ε, τις ουσίες και τα επίπεδα κατόφλια των ουσιών αυτών και αποφασίζει για την ταξινόμηση των επιχειρηματιών. Αν δηλαδή είναι υψηλού κινδύνου ή αν είναι αυξημένου ή υψηλού κινδύνου, είναι μια προσαρμογή στην ισχύουσα οδηγία COP. Τώρα, το πρώτο, οι, τροπολογίες του παρατήματος 1 εμπλέκουν τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις μελλοντικές τροπολογίες του παραρτήματος που έχουν σχέση με τις τεχνολογικές αλλαγές ή κάποιες αλλαγές που αφορούν την ταξινόμηση των επικίνδυνων ουσιών. Ε, η Κομισιόν λοιπόν προτείνει μια, ε, ένα ευρωπαϊκό σύστημα εξαιρέσεων για τις ε, ουσίες και ένα άλλο σύστημα που θα δώσει τη δυνατότητα να εισαχθούν νέες ουσίες στο παράρτημα. Οι τροπολογίες του παραρτήματος 1 θα γίνουν με βάση τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως κατεξουσιοδότηση πράξης. Τέλος, οι τροπολογίες του παρατήματος 1 πρέπει να θεωρηθούν το βασικό στοιχείο της πρότασης. Δεύτερον, στη διαδικασία αναθεώρησης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να εισάγει περιορισμένες ε, ρυθμίσεις, αλλαγές για να ερμηνευθούν και να ενημερωθούν κάποιες διατάξεις χωρίς να γίνουν σε βάθος αλλαγές στο υφιστάμενο σύστημα. Αυτά αφορούν χωρο, χωροταξική διαχείριση, ενημέρωση του κοινού και άλλες αλλαγές όπως προθεσμίες για την αναφορά των ατυχημάτων κλπ. Οι τροπολογίε λοιπόν στο παράρτημα 1 είναι σαφώς το σημαντικότερο στοιχείο τη οδηγία, και όπω σας είπα και πριν, το παράρτημα αυτό προσαρμόζει την οδηγία σύμφωνα με τις διατάξεις του, κανονισμού COB και του πεδίου εφαρμογή του. Ο αριθμό των επιχειρηματιών που δεν ε, ε, δεσμεύονται από τι διατάξει τη οδηγία σε ή που θα συμπεριληφθούν σε αυτή. Αυτό έχει συζητηθεί ήδη στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, στο σεμινάριο που έγινε εκεί. Ο χημικός κλάδος υπονομεύει τους υπολογισμούς. Για μας λοιπόν, εμεί πρέπει να σκεφτόμαστε την διαδικασία που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αλλάζουν αυτά τα παραρτήματα στο μέλλον. Δεν θέλω... Α, η τελική... Δεν θέλω να πω την τελική θέση που θα έχει η γνωμοδότησή μου. Θα ήθελα όμως να ακούσω τους σκιώδεις εισηγητές για να ακούσω και τη δική τους άποψη από αυτού. Όσον αφορά τις υπόλοιπες τροπολογίες, θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά θετικές και εξηγούν πολλά ζητήματα πρέπει να αντιμετωπίσουμε με θετικό τρόπο τις διατάξεις ενημέρωσης του κοινού, την της πρόσβασης σε νομικές διαδικασίες και το θέμα της ενημέρωσης και αναφοράς. Η Κομισιόν ήδη έχει προσδιορίσει τις ε, προθεσμίες για την αναφορά των ατυχημάτων. Θα πρέπει όμως και εμείς να βελτιώσουμε την ποιότητα των αναφορών των ατυχημάτων ε, στο σύστημα. Βασικός στόχος του συστήματος είναι να, ε, καταλήξουμε σε συμπεράσματα και να μάθουμε από την εμπειρία και από τα λάθη των άλλων. Ε, πρέπει λοιπόν η ποιότητα των αναφορών να βελτιωθεί. Δυστυχώς κάποιες αναφορές δεν είναι απόλυτα πλήρης. Αυτή τη στιγμή 25 έως 30, ε, ε, ατυχήματα κάθε χρόνο αναφέρονται και πρόσφατα ο αριθμός των ατυχημάτων μοιάζει ότι περιορίζεται. Η Κομισιόν λοιπόν πρότεινε αλλαγή κατοφλίου για την αναφορά των ατυχημάτων, ώστε να μπορέσουν να συμπεριληφθούν και μικρότερα ατυχήματα και να μάθουμε ακόμα καλύτερα από τα λάθη ο ένας του άλλου. Επίσης θέλω να επανέλθω στο θέμα της ενημέρωσης της κοινή γνώμης του κοινού γιατί το θεωρώ ε, σημαντικό για τη δουλειά της δικής μας Επιτροπής. Είναι σημαντικό οι κοινότητες που είναι κοντά σε επιχειρηματίες σε βέζο να γνωρίζουν τους υφιστάμενους κινδύνους. Δηλαδή, είναι σημαντικό να υπάρξει ευαισθητοποίηση, να ενημερωθούν για την υφιστάμενη απειλή και να γνωρίζουν το είδος του τι πρέπει να κάνουν σε περίπτωση ατυχήματος. Σαφώς σε τέτοιου είδους ε, καταστάσεις βασικό στοιχείο είναι συνεργασία επιχειρηματιών και αρχών και ενημέρωση της κοινή γνώμης του κόσμου για το τι πρέπει να κάνει σε κάθε περίπτωση η μορφή και η μέθοδος μετάδοσης των πληροφοριών είναι και αυτή εξαιρετικά σημαντική, ώστε να μπορέσουν οι πολίτες να μην κατακλείζονται υπερβολικά συχνά από πληροφορίες που καμιά φορά μπορεί να αποδειχθούν και ακατανόητες για αυτούς. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό οι πληροφορίες αυτές να έχουν διαφάνεια, καθαρότητα και είναι σημαντικό οι πολίτες να μπορούν να αποκτούν περισσότερες πληροφορίες εάν το επιθυμούν. Κάτι άλλο που πρέπει να ξεκαθαριστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια είναι η ευθύνη μετάδοσης πληροφοριών στους, στην κοινή γνώμη. Θα γίνει αυτό από τους επιχειρηματίες ή από τις αρμόδιες αρχές. Η προσέγγιση ποικίλει από κράτος μέλος σε κράτος μέλος εδώ. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι οποιαδήποτε νέα υποχρέωση μπορεί να αυξήσει ουσιαστικά το διοικητικό βάρος των επιχειρήσεων και κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στη συζήτηση που έγινε για, την τροπολογία, για τις τροπολογίες του συστήματος Σεβέζο, ακούστηκαν φωνές που ζητούν να αλλάξει η διφυής προσέγγιση ολόκληρο το σύστημα. Δεν νομίζω όμως ότι αυτό είναι επιθυμητή λύση. Η αλλαγή στο σύστημα προκύπτει κυρίως μέσω των αλλαγών του συστήματος ταξινόμησης των ουσιών και όχι λόγω των νέων απειλών ή του αυξημένου αριθμού ε, ατυχημάτων. Θέλω σχετικά να σας υπενθυμίσω ότι το να θεωρείται κάποια επιχείρηση αυξημένου ή υψηλού κινδύνου, αυτό συνεπάγεται ένα ε, μεγαλύτερο κόστος. Πρέπει λοιπόν να εξισορροπήσουμε τις νέες απαιτήσεις για τους επιχειρηματίες, λαμβάνοντας υπόψη ε, φυσικά θέματα παροχής ασφάλειας, που αποτελεί και τον βασικό στόχο της οδηγίας. Αυτό πρέπει να γίνει με τρόπο ώστε το εφιστάμενο επίπεδο ασφάλειας να διατηρηθεί και να αυξηθεί λίγο και να αποφύγουμε ένα περιττό βάρος. Ελπίζω ότι κατάφερα να σας δώσω κάποιες πληροφορίες για την οδηγία σε βέζο. Θα ήθελα όμως να υπενθυμίσω το χρονοδιάγραμμα της γνωμοδότησης σήμερα. Κάνουμε μια πρώτη ανταλλαγή πληροφοριών. Έχουμε χρόνο μέχρι τις 3 Μαΐου. Η γνωμοδότηση θα μεταφραστεί κατόπιν από τις 24 έως 26 Μαΐου θα ε, μελετηθούν οι θα μελετηθεί το σχέδιο γνωμοδότησης και μετά μέχρι τις 21 Ιουνίου το μεσημέρι μπορούν να υποβληθούν τροπολογίες. Θα πρέπει να ψηφίσουμε στην Επιτροπή ΙΜΚΟ στις 12 Ιουλίου και θα θέλαμε να ψηφιστεί η έκθεση τον Οκτώβρη ε, στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και τον ε, ε, Νοέμβρη ε, στην Ολομέλεια. Ζητώ λοιπόν από τους σκιώδει συγιτές να βοηθήσουν και να ε, πούν τις θέσεις τους. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ για την εμπεριστατωμένη σας παρουσίαση η οποία σίγουρα θα ενημέρωσε πολλούς συναδέλφους από μας. Ας δούμε τώρα τι έχουν να πούν οι σκιώδει Eh, Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω την ε, συνάδελφο για τις ε, πληροφορίες της που συμπεριλαμβάνουν φυσικά και το σεμινάριο που μόλις τελείωσε. Και εγώ θα ήθελα να προχωρήσω σε μερικέ γενικές θεωρήσεις για την 9682 οδηγία, δηλαδή τη Σεβέζο 2, η οποία οδηγία θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντική για την μείωση των πιθανοτήτων και των επιπτώσεων των σοβαρών δυστυχημάτων που προκύπτουν από βιομηχανικές δραστηριότητες. Ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι πρέπει να συνεχίσει να προχωρεί σε θέματα ασφάλειας και ότι η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία θα πρέπει να προσαρμόζεται ε, με την ε, νέα ταξινόμηση των επικινδύνων ουσιών. Αυτό πάντα σεβόμενοι το κριτήριο της αποτελεσματικότητας. Θα ήθελα να σταθώ σε, μερικές από τις, ε, σε μερικά σημεία από τις προτάσεις της Κομισιόν. Είναι σημαντικό οι πολίτες, όχι μόνο οι εργαζόμενοι οι οποίοι χειρίζονται αυτές τις ουσίες, όπως έλεγε η συνάδελφη, αλλά οι πολίτες οι οποίοι μπορεί να υποστούν επιπτώσεις να έχουν δυνατότητα πρόσβαση στην πληροφόρηση, συνεχή πληροφόρηση διαφανή και γρήγορη. Να έχουν πρόσβαση στο δίκτυο για να μπορούν να εκμεταλλεύονται ε, τις ανακοινώσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, κυρίως όταν πρόκειται για διασυνοριακά ε, δυστυχήματα. Χαίρομαι που η Κομισιόν ε, θέλει να προχωρήσει σε δημόσιες ακροάσεις και να εμπλέξει και τους πολίτες στη λήψη των αποφάσεων, αλλά θέλω να σταθώ στα εξωτερικά σχέδια κατεπίγουσας ανάγκης. Δεν ξέρω αν θα έπρεπε να έχουμε ένα γενικευμένο σχέδιο για τα κράτη-μέλη ή οι αρμόδιες αρχές του κάθε κράτους μέλους θα ασχολούνται με αυτό το θέμα. Δεύτερο, εγώ έχω μερικές αμφιβολίες για το κατά πόσο θα πρέπει να αφήσουμε την αναθεώρηση του πρώτου παραρτήματος στο μηχανισμό των εξουσιοδοτημένων πράξεων. Και θα ζητούσα, θα παρακαλούσα την Κομισιόν στο εξής. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν πίνακες αντιστοιχίας διότι αυτό το μέσο βοηθάει τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές να ενημερώνονται για το πώς έχει μεταφερθεί σε εθνικό επίπεδο η οδηγία. Σας ευχαριστώ και ελπίζω ότι συνεισέφερα με την τοποθέτησή μου στην έκθεση της συναδέλφου. Ευχαριστώ και εγώ. Η κυρία Παρβάνοβα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ ε, τον εισηγητή, την εισηγήτρια, για την παρουσίασή της και Επίσης, συμφωνώ με τις αλλαγές, τις προτινόμενες αλλαγές. Η ΆΛΔΕ συμφωνεί με την επιβολή αυστηρότερων κριτηρίων ελέγχων. Θα προτείνουμε ορισμένες τροποποιήσεις στις συμπληρωματικές δράσεις Επίσης ε, πυροτεχνικά προϊόντα, ε, παράγωγα πετρελαίου κλπ. θέλουμε να συμπεριληφθούν στον κατάλογο των επικινδύνων ουσιών. Ορισμένα κατόφλια έχουν ε, οριστεί με καθαρά πολιτικά κριτήρια και δεν έχουμε εμπειρικές αποδείξεις που να δικαιολογούν αυτά τα κατόφλια θα προτείνουμε και τροποποιήσεις ε, για μια καλύτερη επισήμανση κινδύνου, ρίσκου, σύμφωνα με το πλαίσιο της νομοθεσίας για το, την προστασία του περιβάλλοντος. Τώρα ο ορισμός μεγάλων ατυχημάτων περιλαμβάνει και κινδύνους με καθυστέρηση εμφάνισης επιπτώσεων. Πρέπει λοιπόν να συμπεριλάβουμε και τις ε, ε, επιπτώσεις στην υγεία με καθυστερημένη εμφάνιση. Ε, να προσέξουμε και το θέμα της επισήμανσης διαφόρων ουσιών που δεν περιλαμβάνονται για τις επικίνδυνες ουσίες που μεταφέρονται υπάρχουν διάφορες ουσίες που δεν περιλαμβάνονται και δεν καλύπτονται, τις οποίες θα θέλουμε εμείς να καλυφθούν και να περιληφθούν. Για τη διαφάνεια προτείνουμε να εξασφαλίσουμε την πλήρη ευθυγράμμιση της νέας οδηγίας με τη σύμβαση του άρχους που έχει συνυπογραφεί από 27 κράτη-μέλη ιδίως όσον αφορά την διαδικασία λήψη αποφάσεων και προσφυγή στη δικαιοσύνη. Θα ήθελα να ζητήσω από την Κομισιόν αν μπορεί να προσφέρει τεχνική βοήθεια ε, στο θέμα των αποζημιώσεων. Όταν δηλαδή σημειωθούν ε, σοβαρά ατυχήματα μπορεί να βοηθήσει οικονομικά στο θέμα των αποζημιώσεων των παθόντων. Ο Πρόεδρος, ε, ποιος άλλος θέλει να μιλήσει. Έντουαρντ, εσύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μία, ένα γενικό σχόλιο μόνο. ελευθερία και ασφάλεια είναι πάντοτε πάρα πολύ πολύτιμες ε, αρχές και πολλές φορές η ασφάλεια και η ελευθερία είναι ε, θύματα ε, κατάχρησης και παραβιάσεων. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από τη Μαλγκορτζάτα να λάβει υπόψη της μία εμπειρία την οποία έχουμε. Στην τελευταία θητεία ε, τσακωθήκαμε αγρίως για την οδηγία REACH. Είχαμε λοιπόν ε, ε, μία οδηγία την οποία συζητήσαμε επί μακρό με πολλούς καυγάδες η οποία τελικά ζημίωσε σημαντικά μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πολλές αναγκάστηκαν να κλείσουν λόγω της οδηγίας REACH. Θα ήθελα λοιπόν να προσέξουμε πάρα πολύ τι ουσίες, τι θα συμπεριλάβουμε, τι θα ζητήσουμε να μην έχουμε το κακό παράδειγμα της Ριτς. Ναι, βεβαίως λέει η κυρία Ρούλε, πρέπει όμως να μελετήσουμε προσεκτικά τις δαπάνες, το τρομερό ατύχημα στην Ουγγαρία με, την κόκκινη, με το κόκκινο ε, χώμα το οποίο βάφτηκε, επίσης το Σοβέτο, τα ξέρουμε όλα αυτά. Να μελετήσουμε λοιπόν τις επιπτώσεις. Είμαι βέβαιος ότι πράγματι ισχύει αυτό. Πρέπει να ενσωματωθεί η ασφάλεια στο σχεδιασμό της διαδικασίας των μονάδων. Αυτό που κάνουμε για τα πρότυπα μπορεί να σχετίζεται με αυτό. Σκέφτομαι την προστιθέμενη αξία που μπορεί να έρθει, να προκύψει από αυτήν την Επιτροπή μας. Πολλά από αυτά που λέμε, θεωρώ, σε σχέση με αυτή την πρόταση, ε, χρησιμοποιούν την προηγούμενη εμπειρία μας και κωδικοποιούμε μια σειρά από βέλτιστες πρακτικές, πρότυπα και διαδικασίες. Οι επιχειρηματίες πρέπει να τα τηρούν όλα αυτά και στο σχεδιασμό αλλά και στη λειτουργία των δραστηριοτήτων τους. Είναι πολύ καλό αυτό υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι ρεαλιστικά αυτά τα πρότυπα και μπορούν να εφαρμοστούν με ενιαίο τρόπο από όλες τις εταιρείες κύριος Κόζοζιτς ε, ε, λέει ότι γίνονται διακρίσεις σε βάρος των μικρών επιχειρήσεων. Ε, αυτό είναι κάτι το οποίο ίσως πρέπει να το κοιτάξουμε. Τώρα, κυρία Βένινγκ, μήπως θέλετε να μας πείτε κι εσείς τι γνωρίζετε επ' αυτού και να σχολιάσετε αυτά που ακούσατε. Thank you, Chair. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ επίσης και την εισηγήτρια και τους σχεώδεις εισηγητές. Είμαστε ιδιαιτέρως ευγνώμονες και ευτυχείς που άρχισε η Επιτροπή σας να δουλεύει σε αυτή την πρόταση της Κομισιόν που όπως πολύ από σας είπατε είναι πολύ σημαντική θέλω για μία ακόμα φορά να υπογραμμίσω αυτό που υπόθηκε. Ο λόγος ε, για τον οποίο ασχολούμαστε με την οδηγία σε Βέζο 2 προκλήθηκε η πρόταση από την ανάγκη να ευθυγραμμιστεί ο ορισμός του πεδίου εφαρμογή ε, της οδηγίας ε, με τους νέους κανονισμούς για τις επικίνδυνες ουσίες που εφαρμόζεται ε, αυτό το ε, παγκόσμιο ε, εναρμονισμένο σύστημα του ΟΗΕ για τις επικίνδυνες χημικές ουσίες. Αυτό αποτελεί το λόγο που επιστρέψαμε σε αυτή την οδηγία σε βέζο. Πρέπει να την ευθυγραμμίσουμε, δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Ως βασι... δεδομένου ότι οι βασικές διατάξεις του σε βέζο παρέμειναν αναλύωτες από τότε που εγκρίθηκε το 1996, φυσικά μας δόθηκε η ευκαιρία να διαπιστώσουμε αν υπάρχουν και άλλες αλλαγές που πρέπει να γίνουν σε αυτή την αλλαγή υπό το φως των εκθέσεων εφαρμογής που έχουμε λάβει εδώ και αρκετό καιρό πια. Ε, το ευχάριστο είναι ότι η ισχύουσα οδηγία έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην μείωση των σοβαρών ατυχημάτων και των συνεπειών τους. Όμως, εξακολουθούμε περίπου κάθε χρόνο να έχουμε 20 έως 35 σοβαρά ατυχήματα τα οποία κοινοποιούνται στην Κομισιόν. Και πρέπει να παραδεχτούμε ότι αυτά είναι πάρα πολλά. Έτσι, στο πλαίσιο αυτό πρέπει να συνεχίσουμε να επιδιώκουμε την περαιτέρω μείωση του κινδύνου τέτοιων ατυχημάτων και εάν συμβούν να περιοριστούν οι συνέπειές τους. Επειδή ενδεχομένως το κόστος ε, τέτοιων ατυχημάτων είναι πολύ ψηλό για την υγεία και τον άνθρωπο και το περιβάλλον όπως είπατε, δεν θα μπορέσουμε μόνο να εξοικονομήσουμε χρήματα για την κοινωνία, αλλά κυρίως να δώσουμε σε κάθε πολίτη την βεβαιότητα ότι το περιβάλλον στο οποίο ζει είναι καλύτερο και ασφαλέστερο. Όπως είπα, η βασική αλλαγή που απαιτείται είναι η ευθυγράμμιση του λεγόμενου παραρτήματος 1 και η διόρθωση του πεδίου εφαρμογή σύμφωνα με το σύστημα ε, ταξινόμησης του COP. Είδαμε σήμερα το απόγευμα στο σεμινάριο ότι η ευθυγράμμιση αυτή δεν είναι απολύτως εύκολη. Χρειάζεται μία σε βάθος ανάλυση των πιθανών εναλλακτικών λύσεων. Τα κριτήρια της Κομισιόν, αφού συζητήθηκαν βεβαίως, έγιναν συζητήσει και με τεχνικούς εμπειρογνώμους εδώ και σχεδόν δύο χρόνια, τα κριτήριά μας λοιπόν για την επιλογή της καλύτερης εναλλακτική ήταν να διατηρηθεί το επίπεδο ε, προστασίας, αλλά ταυτόχρονα να ελαχιστοποιηθούν τυχόν επιπτώσεις στο πεδίο εφαρμογή της οδηγίας. Εμείς θεωρούμε ότι η πρότασή μας επιτυγχάνει αυτή την ισορροπία και επειδή υπάρχουν σχέσεις μεταξύ του Σεβέζο και της χημικής νομοθεσίας, οποιασδήποτε αλλαγές στα πλαίσια της ACP θα επηρεάσουν και την Σεβέζο 3. Αυτός είναι, αυτή είναι η σχέση που υπάρχει και δεν μπορούμε την αλλάξουμε καθώς μελετάμε την οδηγία Σεβέζο 2. Όμως, επειδή το παραδεχόμαστε αυτό, έχουμε συμπεριλάβει στην πρότασή μας και κάποια ευελιξία. Ένα μηχανισμό που επιτρέπει την τον περιορισμό οποιοδήποτε ε, ανεπιθύμητων επιπτώσεων στο μέλλον λόγω των χημικών ουσιών που δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε στο μέλλον την ανάγκη να μπορούμε να αποκλείσουμε ή να συμπεριλάβουμε, εξαρτάται, οι ουσίες από το πεδίο εφαρμογή της ΣΕΒΕΖΟ ανάλογα με το αν και κατά πόσον αποτελούν κίνδυνο για σοβαρό ατύχημα. Άρα, ενώ το εργαλείο, το COP, αποτελεί το βασικό εργαλείο, εξακολουθούμε ε, ε, να θεωρούμε ότι με αυτές τις ρήτρε εξαίρεσης μπορούμε να διατηρήσουμε την απαραίτητη ευελιξία για να μην τιμωρήσουμε με το υφιστάμενο σύστημα, ενώ να συμπεριλάβουμε κάποιες ουσίες που τυχόν δεν έχουμε ακόμα συμπεριλάβει και θα έπρεπε. Πέραν αυτού έχουμε ενημερώσει και ξεκαθαρίσει ή βελτιώσει κάποιες άλλες διατάξεις, όπως αναφέρθηκε εδώ. Μιλάμε συγκεκριμένα για τους τομείς της δημόσιας συμμετοχής, της δημόσιας πρόσβασης στις πληροφορίες, τη πρόσβαση στη δικαιοσύνη και στις επιθεωρήσεις. Θεωρούμε ότι οι απαραίτητες πληροφορίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια και η κατάλληλη συμπεριφορά σε περίπτωση ατυχήματος είναι κάτι που θα πρέπει να είναι άμεσα και πόντοτε διαθέσιμο στο κοινό μέσω του διαδικτύου. Επιπλέον ε, πρέπει να γίνονται δημόσιες διαβουλεύσεις και συγκεκριμένες, ε, έχουν προταθεί συγκεκριμένες διατάξεις πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε περιπτώσεις πολιτών για θέματα που επηρεάζουν την ασφάλειά τους. Τέλος, έχουμε προτείνει ενισχυμένα πρότυπα για τις επιθεωρήσεις συμπεριλαμβανομένων και της συχνότητας που βεβαίως είναι σημαντική για την αποτελεσματική ε, εφαρμογή των κανόνων. Κύριε Πρόεδρε όμως πρέπει να επισημάνω ότι οι αλλαγές αυτές είναι περιορισμένες στο πεδίο εφαρμογή του, στηρίζονται σε αυτό που έχουμε τώρα. Υπό το φως όμως των εκθέσεων που έρχονται από τα κράτη-μέλη για την εφαρμογή έχουμε προσπαθήσει να καλύψουμε τα εμφανή κενά. Λοιπόν, στο σημείο αυτό θα κλείσω όσον αφορά τα όσα λέω εγώ και προσβλέπω σε μια επικοδομητική συζήτηση. Δεν ξέρω εάν θέλετε να ασχοληθώ με ένα από τα δύο, ένα-δύο θεματάκια που ετέθησαν. Δεδομένου ότι έχουμε χρόνο, νομίζω ότι θα ήταν ευπρόσδεκτο, ευχάριστο για τους εισηγητές να σας ακούσουν. Οπότε, θα θέλω να διευκρινίσω το αίτημα που αφορά τα σχέδια εκτάκτου ανάγκης, τι πρέπει να γίνει. Μιλάμε για εξωτερικά σχέδια εκτάκτου ανάγκης. Πρέπει δηλαδή να εκπονηθούν από τις αρμόδιες αρχές, ανάλογα με το πώς βεβαίως έχει στήσει το σύστημά της η χώρα. Θα πρέπει να είναι τοπικές, περιφερειακές ή και εθνικές αρχές. Όσον αφορά τις μικρομεσαίες, πράγματι είχαμε ε, κάποια θέματα προς συζήτηση, ίσως και να παρευρεθήκατε και στο σεμινάριο. Αυτό που διαπιστώσαμε στη διαδικασία αναθεώρησής μας είναι ότι φυσικά υπάρχουν μικρομεσαίες αλλά οι μικρομεσαίες δεν σημαίνει ότι ο κίνδυνος είναι χαμηλότερος. Υπάρχουν αρκετές μικρομεσαίες που αποθηκεύουν εξαιρετικά ε, τοξικές ή έφλεκτες ουσίες και μπορούν να προκαλέσουν ζημιά πολύ μεγαλύτερη από κάποια ε, μεγάλη εταιρεία που αποθηκεύει μεγάλες ουσίες αλλά που εντάσσονται σε λιγότερο τοξική κατηγορία. Πρέπει λοιπόν να το αντιμετωπίσουμε αυτό ε, για λόγους ασφάλειας έχουμε, και το είπα αυτό και στο σεμινάριο, όχι δεν έχουμε πολλές πληροφορίες ε, από τα κράτη-μέλη για τις μικρομεσαίες ως ποσοστό του συνολικού αριθμού των 10.000 εγκαταστάσεων. Ε, ξέρουμε ότι με την πρότασή μας ελάχιστες αλλαγές θα υπάρχουν στην ε, υπάρχουσα ισορροπία στη σχέση μεγάλων επιχειρήσεων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Όσον αφορά τις μικρομεσαίες υπάρχουν και κάποια ζητήματα που αντιμετωπίζουμε όπως παραδείγματος χάρη κάποιες εταιρείες, εάν δεν ανήκουν στην κατηγορία του υψηλού κινδύνου, έχουν και περιορισμένες απαιτήσει. Εξαρτάται όμως πάντα από την κατηγορία κινδύνου στην οποία έχουν ενταχθεί, στο αυξημένου ή του υψηλού, το ανώτατο δηλαδή. Τώρα, για τις μελέτες χρηματοοικονομικής στήριξης πρέπει να πω ότι υποθέτω ότι υπάρχει σχέση με το Risk Facility Fund, νομίζω ονομάζεται. Είναι ένα, αυτό συζητείται σε ένα διαφορετικό πλαίσιο. Δεν θεωρούμε ότι είναι σκόπιμο να αναφερθεί αυτό εδώ, σε αυτό το πλαίσιο, αλλά στο πλαίσιο της διαδικασίας αστικής ευθύνης. Εμείς λοιπόν δεν θεωρούμε ότι αυτά τα θέματα θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε αυτήν εδώ την οδηγία. Το κριτήριο της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας βεβαίως ενδεικτικά έχουμε εντοπίσει ψάχνοντας ουσία προς ουσία κατά την μεταφορά του συστήματος COP στο σύστημα Σεβέζο 3, ότι συνολικά μειώνουμε το πεδίο που καλύπτουν οι εγκαταστάσεις κατά περίπου 2%. Πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχουν 440 περίπου εγκαταστάσεις που βγαίνουν γιατί οι ουσίες τους δεν θεωρούνται πλέον ε, δεν εντύπτουν στις κατηγορίες αυτές που ενέπιταν με το σεβεζο ενω ενώ έχουμε περίπου 220-210 εγκαταστάσεις που τώρα είναι νέες, δηλαδή εμπίπτουν πλέον στην οδηγία ε, για πρώτη φορά. Δηλαδή 184 εγκαταστάσεις φεύγουν συνολικά, αριθμητικά. Θα μείνω εδώ κύριε Πρόεδρε, θα κλείσω και ενδεχομένως κάποια άλλη φορά μπορούμε να συζητήσουμε τα υπόλοιπα. Σας ευχαριστώ Σερμά για την, ε, τις διευκρινήσεις σας. Η κυρία Χάνσλικ ε, σίγουρα θα εξετάσει τις πτυχές εκείνες που θα προσδώσουν περαιτέρω αξίες ε, στην πρόταση της Κομισιόν το, το χρονοδιάγραμμα το έχουμε. Κυρία Χάνσλικ, θέλετε κάτι να προσθέσετε ακόμα. Το μόνο που θέλω να πω είναι να σας ευχαριστήσω για αυτή την επικοδομητική συζήτηση, τις παρατηρήσεις σας. Ευχαριστώ τους και όδους και ευχαριστώ και την Κομισιόν για αυτά που μας είπε σήμερα. Μάσαμε πάρα πολλά και η συμβολή της εκπροσώπου της Κομισιόν θα μας βοηθήσει σαφώς να προσθέσουμε και περαιτέρω αξία σε αυτή τη γνωμοδότηση. Είμαι αισιόδοξη ότι η συνεργασία μας θα είναι Σα Σας ευχαριστώ, ε, δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω. Ευχαριστώ, έχουμε το χρονοδιάγραμμα και <clears throat> μπορούμε να προχωρήσουμε στο τελευταίο ε, θέμα που είναι η... το σχέδιο προπολογισμού 2012. Ε, καλωσορίζω τον κύριο Κόζουτσνικ που είναι εισηγητής και ιδιαίτερα καλωσορίζω τον, την κυρία Φραντσέσκα Μπαλζάνη από την Επιτροπή Προϋπολογισμού που είναι η συγγήτρια η οποία θα μας μιλήσει για το πώς ε, συντίθεται ο προϋπολογισμός, τις διαδικασίες κλπ. Έχουμε επίσης τον κύριο Βάντεκάμπ που είναι η εισηγητής, τον κύριο Μπουζό, τον κύριο Ρόσφορντ, η κυρία Ρίλε, Uh, έχουμε λοιπόν ένα πολύ καλό κύκλο εισηγητών, σκιωδών εισηγητών. Δίνω λοιπόν καταρχά το λόγο στον εισηγητή μας και μετά στην κυρία Παλτσάνη να μας εξηγήσει τις κάπω διαφορετικές διαδικασίες του προπολογισμού, Διαφορετικές από τον προηγούμενο κύκλο προϋπολογισμών θα μιλήσουμε και θα δώσω το λόγο και στους και συνεχεία στον εισηγητή να ολοκληρώσει. Έντουαρντ λοιπόν. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά, διότι μετά από μια σκληρή μέρα εργασίας είναι το τελευταίο θέμα, το οποίο αφορά την τσέπη μας και θα είμαι πολύ γρήγορος. Προσωπικά είμαι ευτυχής που βλέπω ότι η συνάδελφό μας, η κυρία Παλτσάνη, είναι εδώ. Συναντηθήκαμε και την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο και το συζητήσαμε. Αυτό που μου άρεσε στην προσέγγιση της είναι ότι είναι ανοιχτή σε όλε τι προτάσει. Και ε, θέλουμε να διασφαλίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα για ε, τις ε, προθέσει μα. Καλά, υπερβάλλω λιγάκι, αλλά εν πάση περιπτώσει. Θα σας παρουσιάσω καταρχάς ε, το χρονοδιάγραμμα. Το χρονοδιάγραμμα είναι μακρύ, διότι η Επιτροπή Προϋπολογισμού προετοιμάζει μία έκθεση επί της προτάσεως της Κομισιόν και έχουμε όλες τις άλλες γνωμοδοτήσεις. 20 Απριλίου, 20 Απριλίου η Κομισιόν σχέδιο προϋπολογισμό. 23 Απριλίου προθεσμία μεταφράσεων. Η έκθεσή μας θα προετοιμαστεί για τις 14-16 Ιουνίου, μετά ένα μήνα για τροπολογίες, μέχρι 13 Ιουλίου οι τροπολογίες και οι τροπολογίες θα συζητηθούν πριν από τις 31 Αυγούστου και θα ψηφίσουμε στις 31 Αυγούστου. Στην Επιτροπή Προϋπολογισμού η ψηφοφορία θα γίνει τον Οκτώβριο και ελπίζουμε εμείς να ψηφιστεί όλος ο προπολογισμό το Δεκέμβριο. Μία άλλη προθεσμία που μα αφορά οι συζητήσει ε, για τον προπολογισμό καλύπτουν επίση διάφορα πιλωτικά προγράμματα και διάφορε επιτροπέ μπορούν να υποβάλουν αιτήσει Στη δική μας Επιτροπή, την ΙΜΚΟ, θέλουμε το, η μεταρρύθμιση της ενιαίας αγοράς και η εποπτεία της πολιτικής των καταναλωτών. Μπορεί να υποβληθούν και άλλες ιδέες και προτάσεις, οι οποίες πρέπει να έχουν παρουσιαστεί μέχρι τις 3 Ιουνίου. Αυτά θα πω προς το παρόν. Ευχαριστώ. Χαίρομαι ιδιαίτερα που έχετε κάνει όλη αυτή την προπαρασκευαστική εργασία και θέλω να δώσω το λόγο στην κυρία Παλτσάνη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, φέτος, όπως θα, θυμίσει και ο, θα θύμισε και ο Πρόεδρος, θα ήθελα η διαδικασία του προϋπολογισμού να είναι μια διαδικασία ιδιαίτερα σημεριζόμενη από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές. Γιατί ως προς τον ορισμό των τομεακών ε, προτεραιοτήτων, οι αρμόδιες επιτροπές είναι ο ιδανικός χώρος για να ορίσουμε τη στρατηγική του προϋπολογισμού 2012. Η στρατηγική μου πρόταση που εντάσσεται που στο ψήφισμα της 24ης Μαρτίου θέλει να τονίσει ότι αυτή, αυτό είναι, και, είναι η πρώτη χρονιά του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου όπου θέλουμε εμείς να διαμορφώσουμε μία ε, έντονη ευρωπαϊκή διακυβέρνηση. Θέλουμε ένα συντονισμό των εθνικών προϋπολογισμών με τον κοινοτικό προϋπολογισμό για να ορίσουμε τις κοινέ μας προτεραιότητες. Το είπαμε ότι αυτές είναι οι προτεραιότητες της στρατηγικής του 2020 που πρέπει μέσα σε 10 χρόνια να ολοκληρώσουμε. Πρόκειται για μία μέσης διάρκειας περίοδο Πρέπει λοιπόν εμείς να επικυρώσουμε αυτό το στοιχείο του προϋπολογισμού της Ένωσης ότι πρέπει να προσανατολίζει τις επενδύσεις και τις εθνικές πολιτικές ατενίζοντας το μέλλον, ξεπερνώντας δηλαδή το όριο του τρέχοντος οικονομικού έτους. Να βλέπει λοιπόν σε έναν πιο μακρινό ορίζοντα. Πέντε είναι οι στόχοι της ε, στρατηγικής 2020 και το θεμελιώδε σημείο είναι το πρώτο, να ξεκινήσουμε αμέσως, να κάνουμε ένα πρώτο βήμα, να δημιουργήσουμε στην Ευρώπη πιο απασχόληση και μία απασχόληση πιο εξειδικευμένη. Αυτός είναι ο πρώτος στόχος της στρατηγικής 2020. Πρώτος στόχος, ο οποίος συγκεκριμενοποιείται, Άμα ξεκινήσουμε μέσα από ειδικέ επενδύσεις προς την κατεύθυνση της εργασίας, της κατάρτισης, της επαγγελματικής εξειδίκευσης, της υποδομής στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στις ευρωπαϊκές επενδύσεις, εκείνο το κομμάτι της, ε, των υποδομών, κυρίως ενεργειακών υποδομών που από μόνες τους οι χώρες δεν μπορούν να το κάνουν. Λέω λοιπόν ότι θα πρέπει να γίνει αναγνώσιμη πλέον, να, είναι αναγνωρίσιμη στον τωρινό προϋπολογισμό η διαδικασία 2020 οδηγώντας και μία ολοκλήρωση του προϋπολογισμού που θα δίνει νόημα στην ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Θεωρώ ότι αυτό αποτελεί ένα εξαιρετικό μέσο το οποίο το αποκτήσαμε στην Ευρώπη για να καταπολεμήσουμε την κρίση. Μιλάω για τη στρατηγική 2020, αλλά και ένα μέσο για να μπορέσουμε να μετρήσουμε τις δυνατότητες συντονισμού που έχουμε, τους στρατηγικούς μας στόχους, αλλά και ένα εξαιρετικό σύστημα για να εξοικονομήσουμε κονδύλια. Η καινοτομία αυτής της διαδικασίας της φετινής δηλαδή διαδικασίας είναι το να εμπλακούν άμεσα οι επιτροπές, δηλαδή ο προϋπολογισμός να γίνει κάτι το κοινό και να συμβάλλουμε με τις προτεραιότητες μας στο γενικό πλαίσιο του 2020 και να προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα. Το επόμενο βήμα είναι η προθεσμία της 3ης Ιουνίου να στείλουμε ένα προσωρινό κατάλογο των σχεδίων πιλότων και των διαφόρων ε, ερευνητικών σχεδίων. Έχουμε ένα feedback από την Κομισιόν πριν από το Σεπτέμβριο για να παρουσιάσουμε επίσημα μόνο εκείνα τα σχέδια και δράσεις επί των οποίων υπάρχει δυνατότητα συγκεκριμένης ε, ε, δράσης. Η επόμενη προθεσμία είναι μετά το Ιούνιο, είναι η πιο σημαντική. Είναι η φάση εκείνη όπου θα πρέπει να προετοιμάσουμε τις τροπολογίες μας στην πρόταση του Συμβουλίου και να αντιπαρατεθούμε με τους αριθμούς. Να δούμε εάν θα ξεκινήσουμε αμέσως με τον καθορισμό των προτεραιοτήτων επί του προϋπολογισμού, αν θα δώσουμε ένα νόημα στην πολιτική μας δράση, άμα θα δώσουμε αναγνωσιμότητα στη δράση του προϋπολογισμού έτσι όπως θα βγει δηλαδή μετά από το Συμβούλιο. Αυτός είναι ο αποτελεσματικότερος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε τη διαδικασία που και με μία και μόνη διαδικασία και με μία και μόνη συνδιαλλαγή να καταφέρουμε να είμαστε αποτελεσματικοί, να έχουμε ξεκάθαρες ιδέες για το τι θέλουμε και να είμαστε ρεαλιστές. Διότι αυτή είναι και η πρώτη τελευταία χρονιά ε, πριν από το 2013 έχουμε ελάχιστα περιθώρια, έχουμε έναν άκαμπτο προϋπολογισμό. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, να καταλάβουμε πραγματικά τι είναι πρωτεύον, ποιες γραμμές του προϋπολογισμού πρέπει να ενισχύσουμε. Τα περιθώρια είναι πάρα πολύ περιορισμένα. Η Ισούρε εργάζεται για να δει το τι θα γίνει μετά το 2013 και το θέμα των περιθωρίων αφορά όλη μας τη δραστηριότητα και για την προπαρασκευαστική δράση και για τα σχέδια πιλότους. Πρέπει να καταλάβουμε ποιες είναι οι πραγματικές προτεραιότητες στη διαδικασία του προπολογισμού, να έχουμε μια πολύ συγκεκριμένη προσέγγιση. Πέρυσι διδαχθήκαμε από τη μία και μόνη ανάγνωση ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα πραγματιστές και να κάνουμε το πρώτο βήμα προς τη στρατηγική 2020 που θα καταστήσει ευανάγνωστα, ευανάγνωστο συγγνώμη, τους στόχους μας και θα ορίσει και το χνάρι για τον προγραμματισμό της δεκαετίας. Ευχαριστώ για τις σαφέστατες ε, ε, διευκρινήσεις σας. Είμαι σίγουρη ότι η Κομισιόν θα συμμερίζεται την άποψή σας ότι θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στη χρηματοδότηση ορισμένων δράσεων κλειδιών ε, του 2020. Αυτό σίγουρα καλύπτεται από τα, τους μοχλούς της ενιαίας αγοράς, της πράξης ενιαίας αγοράς. Ήδη έχουμε ε, ξεκινήσει ορισμένες προπαρασκευαστικές εργασίες όπως το Φόρουμ της Ενιαίας Αγοράς και άλλες. Ε, ευθυγραμμιζόμαστε λοιπόν με τον τρόπο σκέψης σας. Όσον αφορά τώρα το χρονοδιάγραμμα χειρισμού, πάντοτε υπάρχουν δυσκολίες ολοκλήρωσης του υπολογισμού πριν από την καλοκαιρινή περίοδο και είναι δύσκολο να συγκεράσουμε τις απόψεις διαφόρων επιτροπών και να τις συλλέξουμε δηλαδή καταρχάς πριν από το καλοκαίρι. Αλλά ας προσπαθήσουμε. Για να δούμε καταρχάς οι σκιώδεις Βάντερκαμπ, Γκέπαρντ, Ρούλε, Ροσφόρ και όποιος άλλο, η κυρία Πάρις, κύριο Βάντερκαμπ πρώτο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και εγώ σας ευχαριστώ κυρία Μπαλτζάνη για τις ε, σαφείς ε, για τα σαφή σας σχόλια. Έχω και γραπτά το χρονοδιάγραμμα. Έχω τρία, τρεις ερωτήσεις. Καταρχάς, το ύψος του προπολογισμού. Ορισμένες φορές έχω την εντύπωση ότι από την Επιτροπή Προϋπολογισμού μας δίνουν διαταγές αυτό υπάρχει, αυτά πρέπει να κάνετε, τελεία και παύλα, ούτε περισσότερα θα πάρετε, ούτε λιγότερα. Ε, όπως ξέρουμε, η Επιτροπή Προϋπολογισμών, η Επιτροπή Προϋπολογισμού είναι η μητέρα όλων των, επιτροπών, ε, άρα λοιπόν θέλουμε έτσι μια περισσότερη μητρική αντιμετώπιση. Ε, σήμερα το απόγευμα αναφερθήκατε και στον Επίτροπο κύριο Μπαρνιέ, είχαμε μια εμπεριστατωμένη συζήτηση μαζί του και προκύπτουν ζητήματα προϋπολογισμού. Ωραία είναι το, πράσινο το μπλε αυτό εγχειρίδιο με τους μοχλούς, τους 12, κλειδιά, δράσεις κλπ. Αλλά αυτά όλα συνοδεύονται από χρηματοδοτικά μέσα. Και τρίτον, η προστασία καταναλωτών, όπως ξέρετε, η εσωτερική αγορά μεγαλώνει συνεχώς, διευρύνεται και όλο και περισσότερο θέλουμε να προωθούμε τον τομέα της προστασίας καταναλωτών. Αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει πάντοτε. Υπάρχει, δημιουργούνται προβλήματα. Το 2020 και επειδή είμαι και μέλος στη ΛΥΜΠΕ, μας λένε ότι συνέχεια ότι στο 2020 είναι η απόλυτα οριστική προθεσμία, είναι το ε, σημαντικό ορόσημο. Τι θα γίνει όμως με τις προτεραιότητες του ΙΜΚΟ. Εμείς προσπαθούμε να ευθυγραμμιστούμε προς τα, τους στόχους του 2020 που υποτίθεται ότι είναι το ορόσημο για όλους μας. Τι κάνει όμως ο προπολογισμό. Ο πρόεδρος, ναι, με ενδιαφέρει, με ενδιαφέρει η σχέση μητέρας και τέκνων, έστω και ας είναι σε, σε επίπεδο επιτροπής. ο, ο μιλητής επανέρχεται. Όταν προσπαθώ να εξηγήσω στα παιδιά των γυμνασίων και λυκείων, ε, τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, τους λέω, είναι πρώτα μία ε, κοινότητα ειρήνης και δεύτερον μία εσωτερική αγορά. Αυτά τους λέω. Η κυρία Γκέπαρντ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τους δύο εισηγητές. Κοζούτσνικ και Μπαλζάνη που ε, μας ενημέρωσαν εις βάθος και για το τι ε, θα, θα γίνει στο μέλλον, τι έρχεται κατά πάνω μας. Θέλω πραγματικά να ληφθούν υπόψη σοβαρά οι εργασίες των επιτροπών. Ε, ίσως δεν έχει κυκλοφορήσει τόσο πολύ, δεν έχουν κυκλοφορήσει τα σχόλια γιατί δεν είναι και πολλές επιτροπές ε, παρούσες εδώ. Ε, ίσως η Επιτροπή Προϋπολογισμού να μην έχει ενομοιρωθεί. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η Επιτροπή Προπολογισμού είναι πάρα πολύ σωστό αυτό. Θα πρέπει να συλλειτουργεί με τις άλλες επιτροπές. Προτείνω, κύριοι Κοζούντσνη και Βάντερ Κάμπερ, σε αυτά τα θέματα προτεραιότητας που είχαμε μέχρι τώρα να επιμείνουμε. Δηλαδή να παρουσιάσουμε μία συνέχεια ο κύριος Κουζούσνικ ανέφερε δύο από αυτά τα προγράμματα. Το πρώτο, το φόρουμ της εσωτερικής αγοράς, το οποίο είναι εξαιρετική σημασία για να μπορέσουμε να προβάλλουμε και δημόσια τι σημαίνει εσωτερική αγορά για τους πολίτες και τι προσφέρει η εσωτερική αγορά, τι είναι και τι προσφέρει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 Πρέπει να δούμε πώς θέλουμε να παρουσιάσουμε αυτή την πολιτική. Πολλές, στα πολλά ταξίδια που κάνουμε στα κράτη-μέλη βλέπουμε ότι οι οργανώσεις προστασίας καταναλωτών αντιμετωπίζουν ακόμα με, μεγάλες δυσκολίες ε, στο να ξεκινήσουν τις ε, ενέργειές τους να δημιουργηθούν, να εδρεωθούν και να αρχίσουν να λειτουργούν. Μήπως λοιπόν χρειαζόμαστε ένα πιλωτικό πρόγραμμα, διότι είπατε ότι μπορούμε να προτείνουμε και άλλες πιλωτικές δράσεις. Λοιπόν, ε, σύσταση καταναλωτικών φορέων, οργανισμών, προστασίας καταναλωτών κλπ. Να μια ιδέα. Τώρα, η, πληροφ... εκστρατεία πληροφόρησης του Solvit, ε, αυτή πρέπει να την ενισχύσει και η Κομισιόν. Δεν ε, πρέπει να ζητήσουμε την εργασία που πρέπει να κάνουν τα κράτη-μέλη να την κάνει η Κομισιόν. Όμως ε, πρέπει να ενημερώσουμε τους πολίτες μας ότι υπάρχει το Solvit, ότι προσφέρει λύσεις ιδίω στο θέμα της αναγνώρισης ε, επαγγελματικής κατάρτισης και ότι πρέπει να ενισχύσουμε αυτή την ενημέρωση. Επίσης είναι σημαντικό στο ευρωπαϊκό επίπεδο να διενεργήσουμε μια εκστρατεία ενημέρωσης, έτσι ώστε τα κράτη-μέλη τα οποία δεν λαμβάνουν σοβαρά υπόψη αυτό το πρόγραμμα να αναγκαστούν να το κάνουν. Εάν οι πολίτες πιέσουν, τότε θα αναγκαστούν και ε, οι κυβερνήσεις και οι διοικήσεις, οι εθνικές διοικήσεις να δημιουργήσουν τις απαραίτητες θέσεις. Αυτά είναι τα τρία σημεία που μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα από πλευράς Επιτροπής μας. και περιμένω με πολύ ενδιαφέρον να δω αν προκύψουν και ποιες θα είναι οι συμπληρωματικές προτάσεις. Ευχαριστώ. Πρέπει να συνδέσουμε τα πεπραγμένα με τις νέες διαδικασίες. Ο κύριος Ροσφόρντ. Θα δείτε κύριε Πρόεδρε ότι οι, πιό οι προ... προτεραιότητες της Άλντε είναι πολύ κοντινές και θα εκφραστώ και στο όνομα του κυρίου Μπουζόη. Φυσικά, φυσικά κυρία Μπαρσάνη, ένας προϋπολογισμός θα πρέπει να εξυπηρετεί την ιδέα της ανάκαμψης, την έμονη ιδέα της ευρωπαϊκής ανάκαμψης. Εγώ λέω στον κύριο Τεκάμπτ ότι δεν πρόκειται για θρησκευτικό πρόβλημα, δεν σεβόμαστε εδώ τις ιερές αγελάδες. Απλώς η στρατηγική 2020 είναι μια στρατηγική γύρω από την οποία τα κράτη-μέλη συμφώνησαν. Και ακριβώς επειδή τα κράτη συμφώνησαν, θα πρέπει να τη χρησιμοποιήσουμε ως μοχλό για να είμαστε μέσα σε μια λογική συμβατότητας. Μιλάμε εμείς για το Single Market Act. Ακούσαμε τον Επίτροπο ε, Μπαρνιέ. Για μας αποτελεί ένα στοιχείο ε, απαράβατο για την Επιτροπή μας και θεωρούμε ότι το, το ΣΜΑ πλέον κλείνεται σε, δια, σε διάφορα κεφάλαια που είναι πολύ σημαντικά. Για μας, ας πούμε, η ψηφιακή αγορά, όπου η απασχόληση και ο ανταγωνισμός πρέπει να ενισχυθούν. Μιλάτε για δύο σημεία για το φόρουμ της ενιαίας αγοράς ε, εσείς πρόεδρε νομίζω το αναφέρατε, το 2011 χρηματοδοτήθηκαν και για μας είναι κάτι το πολύ σημαντικό, είναι αυτονόητο το οποίο θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί και το 2012. Και μετά, last but not least, χρειάζεται και μια χρηματοδότηση για την πολιτική των καταναλωτών. Και εδώ χρειαζόμαστε περισσότερα κονδύλια. Ο κύριος Δεκάμπτ ε, εξέτασε και την πιθανότητα ε, για περισσότερο χρήμα. Πρέπει λοιπόν και εμείς να εστιαστούμε γύρω από την πολιτική των καταναλωτών και προγράμματα που έχουν ένα γενικότερο χαρακτήρα για την Ένωση. Η κυρία Ρίλε. Πέρσι, ήμουν εισηγήτρια πέρσι και είχαμε προβλήματα βεβαίως με τις ενώσεις καταναλωτών στην Ανατολική Ευρώπη. Οπότε συμφωνώ ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα, αλλά ταυτόχρονα πρέπει τα κονδύλια να χρησιμοποιηθούν ε, με, με φρόνημα, έτσι, λογική και φρονημάδα. Δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω. Ο Πρόεδρος. Κάτι άλλο που κανείς δεν ανέφερε, την έκθεση του κυρίου Σαλβίνη, τελωνία. Εξυγχρονισμός των τελωνίων. Πολύ σημαντικό θέμα και σημαντικό και στη χρηματοδότησή του από τον προϋπολογισμό. Πρέπει να αντανακλάτε το χρονοδιάγραμμα της έκθεσης με αυτό του προϋπολογισμού. Επίσης, η Κομισιόν κινείται στο θέμα της εποπτείας της λειτουργίας της αγοράς. Έχουμε ε, προβλέψει ορισμένες πιστώσεις ε, που συνδέονται με την πράξη της ενιαίας αγοράς. Ε, δεν θέλουμε να δώσουμε την εντύπωση ότι είμαστε μία ακριβή επιτροπή υπέρ των πολλών εξόδων. Δεν θα, μας, δεν θα αρέσει αυτό στην Επιτροπή Μητέρα. Κυρία Μπαρζάνη, θέλετε να μας συμβουλέχετε κάτι άλλο να μας πείτε, καμία συμβουλή και ο κύριος Κούζισνικ ή ο Ed, τέλο πάντων σήμερα, όλοι τον αποκαλούν Έντβαρτ. Θα ολοκληρώσει. Ευχαριστώ για, αυτά τα πρώτα, για αυτές τις πρώτες προτάσεις που είναι πολύ σημαντικές. Να απαντήσω όμως σε πιο δύο ειδικέ ε, ερωτήσεις για να αξιοποιηθεί, και πιο, να αξιοποιηθεί καλύτερα αυτή η διαδικασία. Ποια είναι τα όρια, ρώτησε κάποιος, ε, για να ε, ορίσουμε εμείς την κοινοβουλευτική μας θέση εναντί του Συμβουλίου. Ε, τα όρια είναι φυσικά τα όρια της σαφήνιας. Πρέπει να είμαστε λοιπόν συγκεκριμένοι, να έχουμε μία πρόταση που θα γίνει δεκτή, γιατί πρέπει να φτάσουμε μετά στη συνδιαλλαγή και μετά τα περιθώρια. Δηλαδή, ποιες είναι τα όρια που έχουμε βάσει των δημοσιονομικών προοπτικών που ισχύει μέχρι το 2013. Αν εμείς από την αρχή έχουμε μία ρεαλιστική αντιμετώπιση, έχουμε περισσότερες δυνατότητες στην συνδιαλλαγή τον επόμενο, το επόμενο φθινόπωρο να καταλήξουμε σε μία συμφωνία. Το θέμα των σχεδίων πιλότος και των προπαρασκευαστικών ε, πράξεων είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό. Στην μεγάλη συζήτηση που είχαμε με την Κομισιόν για να δούμε πώς θα κινηθούμε καλύτερα σε αυτό το πεδίο, διαπιστώσαμε ότι η Κομισιόν δεν θα διαχειρίζεται μόνη της τις, ε, τα σχέδια πιλότους και τα προπαρασκευαστικά σχέδια, διότι αντιμετωπίζει τεχνικά προβλήματα. Πρέπει λοιπόν να είμαστε καινοτόμοι να προσπαθήσουμε με φροντίδα να παρουσιάσουμε προτάσεις οι οποίες δεν καλύπτονται ήδη από άλλα προγράμματα και κυρίως άμα λειτουργήσουν όλα αυτά, άμα λειτουργούν μάλλον τα ισχύοντα, να κοιτάξουμε να τα συνεχίσουμε. Γιατί ένα σχέδιο πιλότος που λειτουργεί καλά από προπαρασκευαστικό σχέδιο μπορεί να μετατραπεί σε πολιτική της Ένωσης. Θα πρέπει λοιπόν εμείς να παρακολουθήσουμε αυτά τα σχέδια πιλότους, τα οποία καταλαβαίνουμε μετά από ένα χρόνο αν λειτουργούν ή όχι. Η κριτική συνέχεια είναι το καλύτερο εργαλείο σε αυτή τη φάση. Μετά υπάρχουν πολλά θέματα που εφήχθησαν και τα οποία είναι της ουσίας και τα οποία θα είναι και πάρα πολύ χρήσιμα για να μπορέσουμε να διαβάσουμε μέσα από το μάτι των προσδοκιών μας την πρόταση της ε, Κομισιόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που ήρθατε στην Επιτροπή μας και περιμένουμε, ε, είμαστε βέβαιοι ότι θα συνεργαστούμε πολύ καλά μαζί σας. Ο Έντβαρντ, ο εισηγητής, θα είμαι πολύ σύντομος για να μην σας καθυστερώ, δεν ζηλεύω τη συνάδελφό μας, την κυρία Παλτζάνη, στο ρόλο της και εκτιμώ ιδιαίτερα που θέλει να περάσει από τις διάφορες επιτροπές, αλλά εγώ πιστεύω η δική μας επιτροπή είναι καλύτερη, διότι είμαστε μία οικογένεια και έχουμε και τη δική μας θρησκεία. Συμφωνώ με την αρχή της συνέχειας βεβαίως και όλα μας τα σχέδια και τα προγράμματα πρέπει να έχουν μια συνέχεια. Δεν είπα ότι ντε και σόνι πρέπει να συμπεριλάβουμε νέα προγράμματα, είπα απλώ ότι υπάρχει δυνατότητα. Εγώ το ρόλο μου τον βλέπω περισσότερο ως ρόλο εισηγητού και θα βοηθήσω οπωσδήποτε την επιτοπή προϋπολογισμού πρέπει να έχουμε μια ενωμένη προσέγγιση ο πρόεδρος. Ωραία, βλέπουμε λοιπόν ε, τι δρόμο πρέπει να ακολουθήσουμε και σύντομα θα έχουμε περισσότερες ε, ιδέες, περισσότερα πιο συγκεκριμένα σχέδια. Σας ευχαριστώ όλους για τη συνεργασία σας και την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε θα είναι τέλος Μαΐου, 24, 25, 26 Μαΐου μακρύ το διάστημα. Έχουμε δύο πράσινες εβδομάδες, έχουμε δύο ομάδες, εβδομάδες ομάδων, έχουμε Πάσχα, Στρασβούργο κλπ. Σας εύχομαι καλό Πάσχα, ελπίζω να ξεκουραστείτε και να είσαστε έτοιμοι για τις ε, σοβαρότατες συζητήσεις που θα κάνουμε στο μέλλον μας. Ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή, ήταν πολύ ε, πυκνή η συνεδρίαση και ευχαριστούμε πάρα πολύ τους διερμηνείς λέει ο Πρόεδρος και εμείς ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ.